Um, Καλημέρα σε όλες και όλους. Έχουμε νομίζω ένα πρώτο πυρήνα για να μπορέσουμε να αρχίσουμε την συνεδρίασή μας, η οποία άλλωστε μεταδίδεται από το διαδίκτυο. Έχουμε μια αίθουσα ασυνήθιστη ας πούμε, είναι αρκετά μεγαλύτερη και δεν βλέπω και καλά καλά τα μέλη. Άλλωστε είναι και πέμπτη πρωί εβδομάδας των ομάδων και πολλοί λείπουν βέβαια σε αποστολές κλπ. Έχουμε ωστόσο ορισμένε σημαντικέ γνωμοδοτήσεις και εκθέσει που πρέπει να συζητήσουμε. Καλώ ήρθατε λοιπόν και έχουμε εκδώσει και τη συνήθι μα έκθεση σχετικά με τι συζητήσει της προηγούμενης εβδομάδα και είναι και δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα μα και έχετε και λάβει αντίγραφα. Τώρα, πριν προχωρήσουμε, να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη για σήμερα. Και είχαμε επιτυχές πέρα των διαπραγματεύσεων για την πρόταση για την ευρωπαϊκή τυποποίηση με το Συμβούλιο την προηγούμενη εβδομάδα και λάβαμε και επίσημη επιστολή από το Συμβούλιο που το επιβεβαιώνει και όπως είδα, είπα ήδη το ίδιο επιτυχή ήταν διαπραγματεύσεις για τον κανονισμό για την ε, πληροφόρηση στην ενιαία αγορά. Θα εγκριθούν επίσημα στην επόμενη συνεδρίασή μας στις 21 Ιουνίου εδώ στην Κοινοβουλευτική μας Επιτροπή και μετά θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην Ολομέλεια, πιθανώς το Σεπτέμβριο, δεν νομίζω νωρίτερα να προλάβουμε θα πρέπει να επανεξεταστούν πρώτα από τις ε, πολιτικές ομάδες, διότι βεβαίως πάντοτε ενδιαφερόμαστε να τηρούμε τις διαδικασίες για συμφωνίες πρώτης αναγνώσεως, προσπαθούμε να κάνουμε όσο γίνεται διαφανέστερες, ώστε να γνωρίζουν οι βουλευτές όλο το κείμενο. 21 έκτου λοιπόν θα υποβληθούν προς έγκριση στην ε, Επιτροπή μας. Τέλος, τα πρακτικά από την 8η Μαΐου τα έχετε στους φακέλους σας και θεωρώ ότι εγκρίνονται μέχρι σήμερα το βράδυ εάν δεν μας υποβάλλετε ενστάσεις. Προχωρώ στο σχέδιο γνωμοδοτήσεως που κάνουμε για λογαριασμό της Επιτροπής Τουρισμού για υπηρεσίες εδάφους στα αεροδρόμια της Ενώσεως. Η συντάκτρια είναι η κυρία Γκάλ Πέλς και η κυρία Ρούλε είναι παρούσα και ο κύριος Κάμπος θέλει να πει κάτι. Αλλά πρώτα η κυρία Γκάλ Πέλς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα θα ήθελα να πω ότι είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη που μπορώ να θέσω υπόψη σας σήμερα το σχέδιο γνωμοδοτήσεως για την ανάκληση της 9667 και κατάργηση δηλαδή της οδηγίας του Συμβουλίου 9667 για τις υπηρεσίες εδάφους στο αεροδρόμιο της Ένωσης. Πρώτα, για ποιο λόγο η Κομισιόν κατέθεσε την πρόταση αυτή. Γνωρίζετε ότι η πρόταση κατετέθη την 1η Δεκεμβρίου 2011, πρόταση δηλαδή νέου κανονισμού για τις υπηρεσίες εδάφους. Το πρόβλημα που σημειώθηκε ήταν ότι η προηγούμενη νομοθεσία που εξακολουθεί να ισχύει και που είχε εγκριθεί το 1996, ε, οι συνθήκες πλαίσια έχουν ε, αλλάξει δραματικά. Διότι πρώτον υπήρξε τεράστια αύξηση αριθμού επιβατών και επομένως υπάρχουν προβλήματα χωρητικότητας. Οι υπηρεσίες εδάφους έχουν γίνει όλο και πιο σημαντικές ως εκ του λόγου τούτου και χρειάστηκε να γίνουν πιο αποτελεσματικές και να βελτιωθεί η ποιότητά τους. Η διαδικασία διαβούλευσης που οργάνωσε η Κομισιόν κατέληξε στο ότι η οδηγία πλαίσιο δεν αρκεί πλέον και έγινε και μία έρευνα με συμμετοχή 27 αεροδρομίων, 67 εταιριών, πολλών αεροπορικών γραμμών, ε, συνδέσμων αεροπορικών γραμμών, ε, αρχών αεροδρομίων και ούτω καθεξής. Έχουμε τα αποτελέσματα της διαβουλεύσεως αυτής και νομίζω ότι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι δι, διτό. Όταν ε, εξετάσει κανείς τις υπηρεσίες εδάφους βλέπει ότι υπάρχουν φραγμοί εισόδου ώστε αυτές οι υπηρεσίες εδάφους δεν είναι αρκετά αποτελεσματικές. Και το άλλο πρόβλημα είναι ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε ευκαμψία, προστασία, προστασία του περιβάλλοντος και όλες αυτές οι πτυχές δεν μπορούν να διασφαλιστούν στα πλαίσια της υφιστάμενης νομοθεσίας. Είναι λοιπόν προς το συμφέρον όλων των πλευρών οι υπηρεσίες εδάφους να είναι Αποδοτικέ, αποτελεσματικέ και για τα αεροδρόμια και για τους επιβάτες. Επίσης θέλουμε να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε με τρόπο ε, αποτελεσματικό όλες τις δυνατότητες που προσφέρουν τα αεροδρόμια και ο κλάδος. Ο κλάδος ανέμενε με μεγάλο ενδιαφέρον τις προτάσεις της Κομισιόν που αποτελούν ένα βήμα προς τα εμπρός και σημαντικό μάλιστα σε σχέση με το παρόν νομοθετικό πλαίσιο. Ωστόσο μένουν ορισμένα θέματα ανοιχτά. Εγώ προσπάθησα να αναλύσω και να ομαδοποιήσω τα ανοιχτά θέματα στο σχέδιο γνωμοδότησής μου και θα ήθελα να τα διεξέλθω μαζί σας. Πρώτο, η απελευθέρωση των υπηρεσιών εδάφου, της αγοράς δηλαδή υπηρεσιών εδάφου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο σχέδιό μου θα δείτε και ελπίζω να συμφωνήσετε ότι η αγορά θα πρέπει να ανοίξει, αλλά με τρόπο ισορροπημένο. Και θα σας πω γιατί. Πρόκειται για ε, επιχειρήσεις εντάσσεως κεφαλαίου με, υψηλά πάγια, με υψηλό πάγιο κόστος και υψηλό ανταγωνισμό. Η Κομισιόν έχει καταθέσει μια πρόταση για τα αεροδρόμια με πάνω από 5 εκατομμύρια επιβάτες ανά έτος και εκεί θέλουν υποχρεωτικά να αυξηθεί ο αριθμός των παρόχων υπηρεσιών από 2 σε 3. Να είναι λοιπόν υποχρεωτικός ο ελάχιστος αυτός αριθμός. Και το έχουν δεχθεί και οι αρμόδιες ε, και ε, οι όμπειροι των επιχειρήσεων. Αλλά θέλω να τονίσω ακόμη ότι κάθε αεροπορική εταιρεία έχει δικαίωμα να κάνει μόνη της εξυπηρέτηση υπηρεσιών εδάφους, εάν το επιθυμεί. Τώρα, εμεί θέλουμε να ενισχύσουμε μια περαιτέρω, ένα περαιτέρω άνοιγμα τη αγορά. Αλλά χωρί να υποστηρίζω εγώ πλήρε άνοιγμα τη αγορά, διότι θα προκαλέσει σημαντικά προβλήματα. Θα μειωθούν οι μισθοί, θα είναι πολύ μεγάλη η πίεση επί των φορέων υπηρεσιών εδάφου, θα χαθεί η ασφάλεια των θέσεων εργασία, θα μειωθούν οι δυνατότητε εκπαίδευση των εργαζομένων, Μπορώ βέβαια να σας αναφέρω πολλά προβλήματα τα οποία θα προκληθούν από ένα ενδεχόμενο πλήρες άνοιγμα της αγοράς. Υπάρχει και ένα μεγάλο θέμα ακόμα, ότι οι χώρες μέλη δηλαδή θέλουν αμοιβαία αναγνώριση των, των αδειών. Όλοι συμφωνούν ότι θέλουν να είναι ελεύθερη διακίνηση μέσα στην ενιαία αγορά. Αυτό είναι σημαντικό. Αυτή ωστόσο η αμοιβαία αναγνώριση των εκκρίσεων λειτουργίας θα πρέπει να βασίζεται σε ανοιχτές ε, διαφανείς διαδικασίες που να μην προκαλούν διακρίσεις, να μην υπάρχουν φραγμοί, να μην υπάρχουν περιορισμοί για να εισέλθει μια επιχείρηση στην αγορά αυτή και επίσης να υπάρχει ελευθερία των επιχειρήσεων να προχωρήσουν σε self-handling εφόσον επιθυμούν. Το άλλο είναι η ευκαμψία, η ευελιξία των, ε, ε, των προμηθειών, των προκηρύξεων εκδηλώσεις ενδιαφέροντος κλπ. Εκεί έχω να πω το εξή. Είπαν οι φορείς ότι χρειάζεται λεπτομερέστερη περιγραφή των διαγωνισμών αυτών και για ουσιώδεις υπηρεσίες κυρίως και η μέγιστη περίοδος επιλογής θα πρέπει να είναι της τάξης των 10 ετών. Εγώ υποστηρίζω την πρόταση αυτή που νομίζω όμως ότι δεν θα πρέπει να περιλάβει μόνο τις ε, Ουσιαστικέ υπηρεσίες, τι ε, σημαντικές υπηρεσίες, αλλά για, θα πρέπει να ισχύσει η δεκαετία για όλες τις υπηρεσίες. Ούτε θα πρέπει να το περιορίσουμε μόνο στο άρθρο 14. Έχω εδώ και μια άλλη πρόταση. Τι θα γίνει εάν μια διαδικασία μειοδοτικού διαγωνισμού δεν είναι επιτυχής και εάν ένας πάροχος υπηρεσιών διακόψει την παροχή υπηρεσιών θα υπάρχει τότε ένα de facto μονοπόλιο. Και σύμφωνα με την πρόταση της Κομισιόν μπορούμε τότε να εκμεταλλευτούμε την δυνατότητα αυτή για να δώσουμε στα αεροδρόμια την δυνατότητα να καθορίσουν τις τιμές για μια χρονική περίοδο. Το τελευταίο μου θέμα είναι για την χρέωση ε, τέλη, δηλαδή για τη χρήση υποδομών. Είναι κάτι σημαντικό που πρέπει να το πούμε επίσης εδώ. Κάθε ένας που χρησιμοποιεί ένα αεροδρόμιο θα πρέπει να μπορεί να έχει ασφάλεια σχεδιασμού, δηλαδή χρειάζονται ε, συγκεντρωτικές, συγκεντρωμένες δηλαδή υπηρεσίες οι οποίες να καθορίζουν τα διάφορα τέλη και εισφορές. Εγώ θα προτείνω εδώ να θεσπιστεί υποχρέωση να δίνεται δηλαδή πληροφόρηση στις εταιρείες και στους παρόχους υπηρεσιών οι δε πληροφορίες αυτές να περιλαμβάνουν και σχεδιο, οποιασδήποτε σχεδιόμενες αλλαγές τιμών ή επενδύσεις και ούτω καθεξής. Αυτές δε οι πληροφορίες να δίνονται υποχρεωτικά σε όλους τους παρόχους υπηρεσιών που ε, δραστηριοποιούνται σε ένα αεροδρόμιο. Και τώρα, οι αρχές των αεροδρομίων θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα να εισπράττουν έξτρα τέλη, τα οποία δεν εισπράττονται διότι έχει κατατεθεί κάποια ένσταση ή έχει ξεκινήσει κάποια άλλη διαδικασία. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν και αναδρομικά να εισπράττουν τα τέλη αυτά οι αρχές αεροδρομίων. Η διαχειριστική αρχή θα πρέπει να παίζει συντονιστικό ρόλο και θα πρέπει να έχει την ε, τις εξουσίες να επιβάλλει κανόνες διοντολογίες, εργατικόδικες διοντολογίες στα, διοντολογίας στα αεροδρόμια. Αυτό είναι το περιεχόμενο της εκθέσεώς μου. Τα ελάχιστα κριτήρια, δηλαδή, εγώ προτείνω για τις υπηρεσίες εδάφους να είναι αυτά, τα, αυτές οι ελάχιστες απαιτήσει δηλαδή, που εναρμονίζονται με τους ε, κοινούς κανόνες της ICAO που έχουν ήδη εγκριθεί από παλαιότερα και λαμβάνουν βέβαια υπόψη και τους κανόνες ασφαλείας και προστασίας των αεροδρομίων και των σχετικών ε, συστημάτων. Αρκούμε σε αυτά κύριε Πρόεδρε και αναμένω να ακούσω τις απόψεις των σκιωδών εισηγητών και των άλλων συναδέλφων μου. Well, thank Ευχαριστώ πολύ για την πλήρη αυτή παρουσίαση για ένα θέμα το οποίο είναι τεχνικό βέβαια, αλλά πολύ σημαντικό θέμα, γι' αυτό είναι σημαντική και η γνωμοδότησή μας. Όλοι μας είμαστε ταξιδιώτες φυσικά και μας ενδιαφέρει. Θα ακούσουμε από τα μέλη και τους σκιώδεις εισηγητές καταρχήν. Η κυρία Σάλτερ Μόζερ είναι παρούσα, δεν ξέρω ο κύριος Μάντελ εδώ, Βίλαντ, Λίουντερς, ο κύριος όχι ακόμα. και η κυρία Εμμάνιουελ Μέρ από την Κομισιόν, από την Γενική Διεύθυνση MOVE που ασχολείται με την εσωτερική αγορά και τα αεροδρόμια. Θα θέλαμε να έχουμε και την απόψη της Κομισιόν γιατί από την Κομισιόν προέρχεται αυτή η πρόταση. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τους σκιώδεις συζητητές. Η κυρία Σάντε Μόζερ έχει το λόγο πρώτα. Σας ευχαριστώ. Συγγνώμη που άργησα. Επειδή όμως είναι ένα τεχνικό θέμα, θα μιλήσω στα δανέζικα. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Θέλω να ευχαριστήσω τον ε, εισηγητή, την εισηγητρία συγκεκριμένα για την έκθεση αυτή. Συμφωνώ για ένα μεγάλο μέρος αυτής της έκθεσης, όχι φυσικά για το σύνολο. Συμφωνώ να πούμε ότι είναι σημαντικό ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι υπηρεσίες εδάφους θα πρέπει να λειτουργούν καλύτερα <clears throat> από ό,τι σήμερα και προσπαθούμε να συμβάλλουμε σε αυτό με μια σειρά τροπολογιών. Θα πρέπει να δούμε κατά πόσο θα πρέπει να τροποποιήσουμε την έμφαση που δίνουμε στη γνωμοδότησή μας ή αν θα πρέπει να συμπληρώσουμε ορισμένες τροποποίησεις. Μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα το να έχουμε κάποια τροποποίηση στη διαδικασία ε, προμηθειών για παροχές εδάφους. Μας ενδιαφέρει καταρχήν να δούμε πώς λειτουργούν οι υπηρεσίες εδάφους για τους ε, επιβάτες ε, και επίσης και για τις αεροπορικές εταιρείες. Εδώ θα πρέπει να καταθέσουμε τροπολογίες προς την κατεύθυνση αυτή. Θα πρέπει οι επιβάτες να περιμένουν να έχουν κάποια πλεονεκτήματα τα οποία θα προκύψουν από τη φιλελευθεροποίηση των υπηρεσιών εδάφους. Χρειάζεται, παραγωγικά, να υπάρχουν ελάχιστα πρότυπα για το χρόνο αναμονής αποσκευών. Είναι πολύ καλό να έχουμε δικαιώματα για τους επιβάτες σε σχέση με την καθυστέρηση των αεροπλάνων, αλλά πρέπει να υπάρξουν και προδιαγραφές σε σχέση με τις αποσκευές. Πρέπει λοιπόν να δούμε τι υπηρεσίες πρέπει να παρέχουν στους ε, Πελάτε του αεροπορικέ εταιρείε και επομένω τι υπηρεσίες πρέπει να υπάρχουν. Επίσης η ιδέα των υπηρεσιών ασφαλείας και αυτό είναι πολύ σημαντικό σε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα με μια υπηρεσία εδάφους θα πρέπει όμως να λάβουμε υπόψη όλα τα στοιχεία που θα μας εξασφαλίσουν ότι αν έχουμε υπεργολαβίε από την ανάδοχο εταιρεία ότι αυτό δεν θα οδηγήσει σε επιδείνωση των συνδικών εργασία των εργαζομένων για θέματα περιβάλλοντος εργασίας ή σε επίπεδο ασφαλείας τους. Πιστεύω ότι βρισκόμαστε όμως στον καλό δρόμο. Θα πρέπει να δούμε αν μπορούμε να βελτιώσουμε τα πράγματα και να εξασφαλίσουμε ότι οι επιβάτες μπορούν να ευνοηθούν από αυτή τη φιλελευθεροποίηση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν σας βλέπω πολύ καλά από εδώ, αλλά ευτυχώς έχω τα γυαλιά μου. Ε, ο κύριος Παπανόβα μου ζήτησε να πω κάποια λόγια για αυτή την έκθεση και θα σας διαβάσω τα σχόλια. Θέλει να συγχαρεί την εισηγήτρια για την εργασία της ε, που κατέληξε σε, μια πολύ ε, σε ένα πολύ ισορροπημένο σχέδιο έκθεσης. Εμείς ως ομάδα υποστηρίζουμε τις προτινόμενες αλλαγές που υποστηρίζουν το περαιτέρω άνοιγμα των υπηρεσιών εδάφους σύμφωνα με την πρόταση της Κομισιόν καθώς και όσον αφορά τις αλλαγές ε, που ε, παρέχουν διασφαλίσεις ε, στην οδηγία. Ο κύριος Παγανόβα πιστεύει ότι θα πρέπει να ενημερωθεί το κείμενο ώστε να αντικατοπτρίζει τις εξελίξεις του τομέα μεταφορών μετά από την έγκριση και την υιοθέτηση της οδηγίας 96-67 και κυρίως όσα αφορά το code sharing, τις πτήσεις κοινού κωδικού Όσον αφορά τις χρήσεις αεροδρομίων, η κυρία Παπανόβα θα ήθελε να δηλώσει ότι υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις υπηρεσίες εδάφους ώστε να καλύπτουν τις προσδοκίες των πελατών. Για αυτό τον λόγο θα πρέπει να εξετάσουμε το δεχόμενο της ενεργού συμμετοχής τους στην επιλογή παρόχων όταν ο αριθμός είναι περιορισμένος καθώς και στον καθορισμό των κωδικών διεντιολογίων. Θεωρεί επίσης ότι τα πρότυπα είναι απαραίτητα ώστε να διασφαλίζεται ότι εν τέλει προστατεύονται τα συμφέροντα των επιβατών. Θα ήθελα εγώ να προσθέσω κάτι προσωπικά, μια προσωπική μου ιδέα. Πολλά ε, αποσκευές ε, χάνονται και καλό θα ήταν να το εξυγχρονίσουμε, να εξυγχρονίσουμε και αυτή την πτυχή αυτοκόλλητα που μπαίνουν πάνω στις αποσκευέ, ε, καθώς και στην κάρτα επιβίβασης ε, να υπάρχει κάποια ένδειξη ταυτότητας, ένα τσίπ ώστε ε, να μπορούμε να εντοπίσουμε και τα δύο ώστε κανείς να μην μπορεί να κλέψει τις αποσκευέ των επιβατών. Είναι μια ιδέα, καλό θα ήταν να το σκεφτούμε. Ευχαριστώ. Η κυρία Ρούλα. Ευχαριστώ. Επανέρχομαι σε αυτό που είπε ο συνάδελφός μου μόλις τώρα για την απώλεια αποσκευών μετά από την πρόταση αυτή που έλαβα της Κομισιόν δηλαδή πήγα και είδα στο αεροδρόμιο Στουτγάρδης που είναι το περιφερειακό μας αεροδρόμιο και μίλησα και με τους αρμόδιους και μάλιστα και με τους εργαζομένους εκεί μαζί με την κυρία Κέπχαρτ μάλιστα πήγαμε και αυτό που μου φαίνεται ότι λείπει από την πρόταση της Κομισιόν και που πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι η αφετηρία στην πραγματικότητα θα έπρεπε να είναι πολύ περισσότερο η τήρηση των προδιαγραφών ποιότητας. Γιατί δεν είναι μόνο η ποιότητα, είναι και η ασφάλεια. Και θα έπρεπε εδώ στη δική μας Επιτροπή, που είμαστε και Επιτροπή Προστασίας των Καταναλωτών, αυτά τα θέματα να παίξουν κέριο ρόλο. Όταν όμως μιλούμε για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τα στάνταρτ ποιότητας και ασφάλειας, δεν είναι δυνατόν να γίνει χωρίς να δούμε πρώτα, να κοιτάξουμε πρώτα ποιες είναι οι συνθήκες εργασίας, οι οποίες έχουν επιδεινωθεί τελευταία και μάλιστα δραματικά. Γι' αυτό πιστεύω ότι μια παραπέρα απελευθέρωση όπως την προτείνει η Κομισιόν θα οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερη επιδείνωση των συνθήκων εργασίας και άρα και σε μείωση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών. Και γι' αυτό είμαι αντίθετη με την πρόταση της Κομισιόν και ευχαριστώ την εισηγήτρια που έχει προβήσει ορισμένε βελτιώσει και αυτέ είναι καταρχήν καλέ, αλλά παρόλα αυτά εγώ πιστεύω ότι ο στόχος, ο πρωταρχικός στόχος των προτάσεων της Κομισιόν είναι εσφαλμένος. Και θεωρώ ότι είναι προβληματική η προσπάθεια να ανοίξει στους υπεργολάβους η αγορά, χωρίς αυστηρά κριτήρια διότι αυτό θα οδηγήσει σε επιδείνωση των προσφερόμενων υπηρεσιών σε όλου του ε, επιβάτε. και βεβαίω και σε επιδείνωση των συνθήκων εργασία. Τονίζω ακόμα επίση ότι είναι απο, απολύτως αμφιλεγόμενο ότι δήθεν ο κλάδο είναι υπέρ. Υπάρχουν πολλοί διαχειριστέ αεροδρομίων οι οποίοι είναι αντίθετοι. Τα συνδικάτα των εργαζομένων επίση είναι αντίθετα. Υπάρχουν και πολλέ αντιστάσει και στι εθνικέ βουλέ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μπίλα. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα επίσης να πω δύο λόγια για να ευχαριστήσω την κυρία εισηγήτρια για αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης. Πιστεύω ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι πολύ σημαντική για τις υπηρεσίες εδάφους και τη μεταρρυθμίσή τους. Πιστεύω ωστόσο ότι η Επιτροπή μας θα πρέπει να επικεντρωθεί στο πώς μέσω αυτής της γνωμοδότησης θα ε, προσφέρει προστιθέμενη αξία για τους ταξιδιώτες για παράδειγμα ο ελάχιστος αριθμός παρόχων ορισμένων υπηρεσιών εδάφους όπως μεταφορά αποσκευών πρέπει να περιοριστεί από δύο σε τρεις παρόχους ε, και μάλιστα ανεξάρτητες ε, υπηρεσίες εδάφους που παρέχονται από αερομεταφόρες. Πιστεύω ότι το ζήτημα του τρίτου παροχού είναι ένας τρόπος να προχωρήσουμε μπροστά και πιστεύω θα επηρεάσει την ευρωπαϊκή αγορά. Πιστεύω δεν πρέπει να υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά τους παρόχους υπηρεσιών εδάφους. Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε το ενδεχόμενο ενός τέταρτου παρόχου για τα μεγαλύτερα αεροδρόμια ε, που υπερβαίνουν μια συγκεκριμένη χωρητικότητα. Ένα πράγμα με το οποίο δεν συμφωνώ είναι ότι αν ανοίξουμε την αγορά των υπηρεσιών εδάφους αυτό μπορεί να παραβιάσει ορισμένες συνθήκες σταθερότητας και μπορεί να διώξει ορισμένους από την αγορά. Πιστεύω ότι η απελευθέρωση της αγοράς θα πρέπει να έχει οικονομικά ωφέλη τόσο για, τις, για τους αερομεταφορείς όσο και για τους καταναλωτές, τους επιβάτες. Αν κοιτάξουμε χώρες όπως οι Ηνωμένε Πολιτείε και η Ιαπωνία Εκεί ο τομέας είναι απολύτως ελεύθερος. Αυτό συμβαίνει και σε ορισμένα αεροδρόμια ήδη της Ευρώπης και πιστεύω ότι δεν πρέπει να επιβάλλουμε περιορισμούς. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες που αφορούν την Επιτροπή Μεταφορών, αλλά έχουμε στοιχεία που μας λένε καθαρά ότι οι τιμές που πληρώνουν οι αερομεταφορείς για τις υπηρεσίες αυτές είναι πολύ υψηλέ και οι, οι διαφορές ε, προκύπτουν από το γεγονός ότι η πρόσβαση για τους μεμονωμένους παρόχους ε, είναι διαφορετική. Πιστεύω λοιπόν ότι εν αυτή η τιμή μεταφράζεται εν τέλει στην τιμή που πληρώνουμε εμείς οι καταναλωτές. Πιστεύω ότι αν απελευθερωθούν οι υπηρεσίες, η ποιότητα των υπηρεσιών θα αυξηθεί και όχι το αντίθετο παρότι μερικοί το ισχυρίζονται και σίγουρα υποστηρίζω και εδώ συμφωνώ με την εισηγήτρια ότι θα πρέπει να εισαχθούν ελάχιστα πρότυπα ώστε να ενισχύθει το συνολικό επίπεδο υπηρεσιών που παρέχονται στα αεροδρόμια. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Γκέπαρντ. Ευχαριστώ. Συμφωνώ. Θα συνεχίσω σε αυτά που είπε η κυρία Ρούλε και εγώ βλέπω ότι είναι πολύ προβληματική η πρόταση της Κομισιόν και εγώ θεωρώ ότι επιπλέον δεν φέρνει καμία προσθέμενη αξία αυτή η πρόταση και ιδίως πρέπει να σταθούμε στο θέμα των εργαζομένων στις υπηρεσίες αυτές γιατί βρίσκονται σε μια κατάσταση όπου έχουν μειωθεί σε σημαντικό βαθμό η προστασία τους και, τα, και η ικανοποίηση των ετοιμάτων τους και πρέπει να λάβουμε υπόψη και αυτή την πτυχή. Επίσης, όταν σε ένα ρομποδρόμιο έχουμε δύο ή τρεις ή τέσσερις ακόμα εταιρείε παρόχων οι οποίες απασχολούν εργαζόμενους, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι επιχειρήσεις αυτές χρειάζονται να έχουν μια υποδομή, να έχουν ένα εξοπλισμό για να μπορέσουν να κάνουν τη δουλειά τους. Αυτός ο εξοπλισμός όμως θα πρέπει να την χάνει συντήρησης για, τα, για να μπορούν να έχουν την υπηρεσία τους στα αεροδρόμια. Όταν έχουμε τώρα πάρα πολλές εταιρείε οι οποίες συνοστίζονται για να παρέχουν αυτές οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης, αυτό μπορεί να είναι πρόβλημα. Το να έχουμε λοιπόν δύο ή τέσσερις ή έξι υποδομές εξυπηρέτησης, αυτό δεν θα κάνει φτηνότερη την εξυπηρέτηση για τους καταναλωτές. Επίσης, δεν μπορώ να φανταστώ ότι η ποιότητα της υπηρεσίας θα βελτιωθεί όταν έχουμε συγχρόνως διάφορες ε, διάφορους φορείς οι οποίοι θα προσπαθούν να εξασφαλίσουν ότι το δικό τους αεροπλάνο θα, για την καθεμία θα είναι το πρώτο που θα εξυπηρετηθεί. Αυτό τελικά νομίζω θα οδηγήσει σε μια χαοτική κατάσταση. <clears throat> θα έχουμε περισσότερες βαλίτσες οι οποίες θα χάνονται από ό,τι από τη τώρα. Νομίζω λοιπόν στον τομέα αυτό δεν είναι καλή ιδέα να προωθήσουμε υπερβολικά τη φιλελευθερωποίηση. Οι υπηρεσίες εδάφους λοιπόν πρέπει να γίνονται με διάφανες διαδικασίες διαγωνισμού, να μην γίνεται με ανάθεση και μόνο, <clears throat> αλλά αυτό μπορεί να οδηγήσει και στο να μην υπάρχει κανένας ανάλογος. Τέλος, μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα το θέμα της ασφάλειας. Όλο περισσότεροι είναι αυτοί οι οποίοι εργάζονται στα αεροδρόμια και όλοι αυτοί οι άνθρωποι, ακόμα και αν ανήκουν σε υπεργολαβικές εταιρείες, θα πρέπει να περνάνε από έλεγχο δεν πρέπει να ελέγχουμε μοναχά τους επι, επιβάτες στα αεροπλάνα, πρέπει να ελέγχουμε και τους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται στα αεροδρόμια και αυτό προσθέτει στο κόστος του όλου εγχείρηματος. Πραγματικά δεν ξέρω. Λοιπόν, αν θα εξοικονομήσουμε κάπου χρήματα και αν θα δώσουμε καλύτερη υπηρεσία στον καταναλωτή. Νομίζω ότι απλώς θα καταλήξουμε σε μια κατάσταση η οποία θα είναι αδιαφανής, θα είναι πολυδάπανη και τελικά δεν πρόκειται να εξυπηρετήσει κανένα ο Ντένις, ο οποίος έχει μόλις έρθει ως σκιοδησίτης. Θες να πεις και εσύ κάτι. <clears throat> Κάποιος άλλος θέλει να πει κάτι και μετά φυσικά και η Κομισιόν θα λάβει το λόγο. Ο Ντένις πρώτα. Ευχαριστώ Μάλκολμ. Εγώ άκουσα μονάχα τα τελευταία λόγια της κυρίας Γκέπχαρτ. Χαίρομαι που άκουσα όμως αυτά γιατί συμφωνώ απόλυτα μαζί της την προηγούμενη εβδομάδα ήμουνα στο Ζάβεντεμ για να δω πώς λειτουργούν οι υπηρεσίες εδάφους στην πράξη. Είναι χρήσιμο να έχουμε μια ίδια εντύπωση για την κατάσταση εκεί. Οι επιχειρήσεις οι οποίες εργάζονται εκεί, είναι δύο αυτή τη στιγμή και μου είπαν ότι πολλές φορές μπορούν, μπορεί να προκύψουν προβλήματα για τις υπηρεσίες που παρέχει το αεροδρόμιο. Δεν θέλουμε να έχουμε λοιπόν μια τρίτη εταιρεία η οποία θα μας ανταγωνίζεται και το Ζάβεντεν προφανώς ξεπερνάει τα 5 εκατομμύρια επιβατών το χρόνο. Θεωρούν λοιπόν ότι δεν υπάρχει χώρος πραγματικά στο αεροδρόμιο για να εγκατασταθεί μια τρίτη εταιρεία εδάφους, ε, υπηρεσιών εδάφους. Θα πρέπει να έχουμε νέες υποδομές για τις αποσκευές για να μπορέσει να υπάρχει μια τρίτη εταιρεία. Νομίζω ότι η Εύλιν Γκέμπχαρτ έχει την ίδια εντύπωση με μένα. Αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει καταρχήν να δούμε αν προκύπτει κάποια προσθέμενη αξία από αυτή την πρόταση και εγώ προσωπικά είμαι σκεπτικιστή σχετικά. Εντυπωσιάζομαι από τον ζήλο των συναδέλφων που κάνανε επιτόπιες έρευνες για τα θέματα αυτά. Η κυρία Ρούλε, η κυρία Γκέμπχαρτ, ο κύριος Δε Γιόγκ έχουν επισκεφθεί διάφορα αεροδρόμια, βέβαια μέσα στα πλαίσια των ταξιδιών του φαντάζομαι, αλλά αυτό δείχνει τη σημασία που αποδίδει η Επιτροπή μα σε αυτή την πρόταση. Αν δεν θέλει κανένα άλλο να λάβει το λόγο, θα ζητήσω από την Κομισιόν να απαντήσει, γιατί βλέπετε ότι υπάρχει κάποιο σκεπτικισμό για την αξία τη πρόταση αυτή. Και σα ε, υπενθυμίζω τη γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου του Λουξεμβούργου που λέει ότι η οδηγία αυτή ότι έχουν αυξηθεί οι υπηρεσίες εδάφους, έχουν μειωθεί το κόστος της εξυπηρέτησης και σύμφωνα με την Κομισιόν έχει αυξηθεί η ποιότητα. Εμείς δεν έχουμε δει ακριβώς την ε, έκθεση αντικτύπου της Κομισιόν. Ίσως μπορούμε όμως να, σταθούμε, να σταθείτε εσείς σε κάποια από τα σχόλια των συναδέλφων. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, κύριε Εισηγήτρια, κυρίε και κύριοι βουλευτές, ε, κυρίε και κύριοι. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Εκπροσωπώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια για το έργο της μέχρι στιγμής ε, που έχει ως στόχο τη βελτίωση της πρότασης της Κομισιόν καθώς επίσης ε, όπως ακριβώς έκανε και το Συμβούλιο στη γενική του προσέγγιση της 22ης Μαρτίου τηρώντας ε, και προσέχοντας ταυτόχρονα τις ισορροπίες, ε, τις υφιστάμενες ισορροπίες κυρίως όσον αφορά το άνοιγμα της αγοράς, των διασφαλίσεων για τους εργαζομένους και κυρίως την ποιότητα των υπηρεσιών για τους επιβάτες. Είμαστε επίση ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που η Επιτροπή, η δική σα Επιτροπή για αυτό το φάκελο. Έχετε τεράστια εμπειρία σε θέματα εσωτερική αγορα και προστασια των Καταναλωτών αναλαμβάνει να γνωμοδοτήσει για αυτό το φάκελο. Έχετε τεράστια εμπειρία σε θέματα εσωτερικη αγοράς ε, πέραν των μεταφορών. Αυτή η οδηγία ε, υπηρεσιών εδάφους ε, βρέθηκε στο επίκεντρο της εσωτερικής αγοράς για την αεροπλοεία. Πριν από 20 χρόνια ακριβώς, οι προκατοχοί μα δημιούργησαν την εσωτερική αγορά ναυσιπλοεία, παρέχοντα στου αερομεταφορείς τη δυνατότητα να καλύψουν τις ανάγκες των επιβατών και να ανοίξουν νέες ε, οδούς ε, ως, χωρίς περιορισμούς όσον αφορά τη χωρητικότητα και τη συχνότητα. Χωρίς αυτήν την οδηγία για τις υπηρεσίες εδάφους το αποτέλεσμα αυτής της εσωτερικής ε, αγοράς ναυσιπλοείας για 500 εκατομμύρια επιβάτες ε, τεράστιους αερομεταφορείς και τεράστια αεροδρόμια όλη αυτή η βιομηχανία δεν θα είχε μπορέσει να δημιουργηθεί. Αυτή η οδηγία ήδη εξ αρχής ε, σεβόταν ιδιαίτερα ορισμένους παράγοντες. Οι υπηρεσίες εδάφους άνοιξαν στην πλειοψηφία τους, στη μεγάλη τους πλειοψηφία σήμερα είναι ανοιχτές στον ανταγωνισμό εκτός από τέσσερις κατηγορίες. Σε αυτές τις τέσσερις κατηγορίες ο Ευρωπαίος νομοθέτης αποφάσισε να διατηρήσουν τα κράτη-μέλη τη δυνατότητα να περιορίσουν τον ανταγωνισμό σε δύο παρόχους με ορισμένες διασφαλίσεις, δηλαδή ότι οι υπηρεσίες εδάφους πρέπει να είναι ανεξάρτητες είτε από το αεροδρόμιο είτε από τον κύριο αερομεταφορέα του αεροδρομίου. 16 χρόνια μετά από αυτή την πρόταση, εμείς προτείνουμε να την επανεξετάσουμε, στο να βελτιώσουμε την ε, αποδοτικότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών. Η αποδοτικότητα σημαίνει να παρέχουμε περισσότερες επιλογές ε, στις αερομεταφορείς για αυτούς τους τέσσερις τομείς υπηρεσιών που εξακολουθούν να ε, ε, υπόκεινται σε περιορισμούς ανταγωνισμού. Δεν σημαίνει ωστόσο απόλυτη επιλογή. Το, κράτο μέλ, το κράτος μέλος θα μπορεί να αποφασίζει και φροντίσαμε να διατηρήσουμε την επιλογή για το κράτος μέλος να μπορεί να αποφασίσει στα μεγάλα αεροδρόμια τα οποία δείχνουν, άνω των 5 εκατομμύριων επιβατών το έτος ο ελάχιστος αριθμός ε, ζητάμε να μην είναι 2 αλλά 3 δεν ζητάμε λοιπόν πλήρη ανταγωνισμό ζητάμε λίγο μεγαλύτερη επιλογή για να αναφερθώ σε ένα σημείο που αναφέρθηκε στη συζήτηση καθίσταται σαφές ότι αν υπήρχαν φόβοι όσον αφορά θέματα χώρου που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και την προστασία, το κράτος μέλος μπορεί να ζητήσει εξαίρεση, μπορεί να το πράξει σήμερα και θα εξακολουθεί να μπορεί να το πράξει και αύριο. Μιλάμε για ένα άνοιγμα λίγο μεγαλύτερο ώστε οι αερομεταφορείς να έχουν λίγο περισσότερες επιλογές ε, όσον αφορά τις υπηρεσίες εδάφους που τους προσφέρουν τα αεροδρόμια. Επιθυμούμε οι συνθήκες ανταγωνισμού να είναι πιο δίκαιες μεταξύ των διαφόρων παρόχων. Αυτή τη στιγμή ε, αερολιμενικοί διαχείριστες ε, έχουν θηγατρικές ε, για τις υπηρεσίες εδάφους και έχουν την τάση να ευνοούν τις δικές τους υπηρεσίες εις βάρος ανεξαρτήτων επιχειρήσεων που προσπαθούν να εισέλθουν σε αυτή την αγορά και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους αερομεταφορείς προσφέροντας ε, ταυτόχρονα καλύτερες ε, μισθολογικές συνθήκες στους εργαζομένους τους. Είναι λοιπόν εξαιρετικά σημαντικό βάσει των όσων είπαμε οι ενδιαφερόμενοι και έχουμε λάβει πάνω από 100 σχόλια να ενισχύσουμε τις συνθήκες ανταγωνισμού ώστε να επιτύχουμε πιο αποδοτική εξυπηρέτηση όσον αφορά την ποιότητα. Συμφωνούμε με τις παρατηρήσεις που ακούστηκαν σε σχέση με τα ελάχιστα πρότυπα ποιότητας. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να καθοριστούν τέτοιου είδους ελάχιστα πρότυπα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για παράδειγμα, επιχειρησιακή απόδοση χρόνος αναμονής ε, για τους επιβάτες ε, στο check-in. Χρόνος παραλαβής αποσκευών. Η πρώτη αποσκευή που φτάνει στον Ιμάντα και η τελευταία αποσκευή που φτάνει στον Ιμάντα παραλαβής. Ε, πιστεύουμε λοιπόν ότι αυτό το στοιχείο της ποιότητας είναι εξαιρετικά σημαντικό και θα πρέπει να ορίσουμε έναν πίνακα στοιχείων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθορίζοντας αυτά τα πρότυπα ποιοτητα. Αυτή τη στιγμή διαφωνούμε με το Συμβούλιο για αυτό το ζήτημα. Το Συμβούλιο θεωρεί ότι αυτό πρέπει να πραγματοποιείται σε επίπεδο αεροδρομίου, κάθε αεροδρομίου ξεχωριστά, Γεγονό που παρουσιάζει ένα κίνδυνο ποικιλομορφία των κριτηρίων μεταξύ αεροδρομίων και ενδεχομένω φραγμό, νέο φραγμό για τους νέους ερχόμενους, τους ανεξάρτητους νέους ερχόμενους ε, φορείς παροχής υπηρεσιών εδάφους οι οποίοι θα δυσκολεύονται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Επίσης, ε, επιθυμούμε να παρέχουμε στα κράτη-μέλη που το επιθυμούν τη δυνατότητα να ενισχύσουν τις διασφαλίσεις του προσωπικού που εργάζεται στις υπηρεσίες εδάφους. Γι' αυτό το λόγο οι διατάξει μεταφορά προσωπικού, μετάταξη προσωπικού είναι εξαιρετικά σημαντικέ. Εάν αύριο ένα κράτο μέλο επιθυμεί να εισάγει διατάξει ώστε το προσωπικό μια επιχείρηση υπηρεσιών εδάφου που εγκαταλείπει την αγορά να επαναπροσληφθεί από μια επιχείρηση υπηρεσιών εδάφους που ε, πήρε τη θέση της, ε, το μεριδιό της στην αγορά. Αυτή η δυνατότητα θα πρέπει να υπάρχει για το κράτος μέλος. Χρειάζεται ωστόσο νομική σαφήνεια για αυτό το ζήτημα. Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος προσφυγών και υπάρχει κίνδυνος κατ' τέτοιο να πραγματοποιηθεί εις βάρος των υπαλλήλων των υπηρεσιών εδάφους. Έχουμε κάποια τεχνική κάποιες τεχνικές παρατηρήσεις όσον αφορά τις τροπολογίες που πρότεινε η συγγήτρια και θα σας ε, στείλουμε αυτές τις ε, τεχνικές φύσεως παρατηρήσεις ε, απευθείας στην συγγήτρια. Θα ήθελα να αναφέρω ένα τελευταίο σημείο που θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό. Τα ζητήματα των υπεργολαβίων και τα ζητήματα του καθορισμού της εξυπηρέτησης διειδίων πόρων. Καλό τα μέλη του Κοινοβουλίου να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά όσον αφορά τους ορισμούς που προτείνει η Κομισιόν. Διότι πέραν ενό τεχνικού ορισμού της εξυπηρέτησης διειδίων πόρων, του self-handling δηλαδή, και του ορισμού της υπερκολαβίας, έχουμε πραγματικά πράγματα που διακυβεύονται με άμεσες επιπτώσεις για τα διάφορα κοινοτικά αεροδρόμια όσον αφορά τον ανταγωνισμό μεταξύ του αεροδρομίου που διαθέτει θηγατρική υπηρεσιών εδάφου, του ανεξάρτητου παρόχου και πραγματικές επιπτώσεις για τους αερομεταφορείς. Συμφωνούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο με τις τροπολογίες της εισηγήτριας η οποία ε, δείχνει ιδιαίτερη προσοχή και σωστά πράττει για όλα αυτά τα ζητήματα του self-handling και τη υπεργολαβίας. Ευχαριστώ. Well, thank you Ευχαριστώ για τις ε, πολύτιμες πληροφορίες που μας δώσατε. Πιστεύω θα ακολουθήσει και μία νέα συζήτηση για το θέμα αυτό στην Επιτροπή Μεταφορών. Κάποιες πάντως από τις ε, θέσεις για τα πρότυπα εξυπηρέτησης θα συζητηθούν και στην επόμενη συζήτησή μας για τα δικαιώματα των ε, επιβατών, όπου έχουμε μια έκθεση πρωτοβουλίας από την Επιτροπή Μεταφορών και μακροχρόνια θα υπάρξουν περαιτέρω εξελίξεις σε τεχνολογικό επίπεδο. Επομένως θα πρέπει να προωθήσουμε τις ε, επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες για τη βελτίωση του επίπεδου υπηρεσιών και ελπίζω ότι και οι συνάδελφοι θα αντιμετωπίσουν το θέμα αυτό. Κυρία Γκαλκέοντς, θέλετε να κάνετε κάποια καταληκτικά σχόλια και να μας πείτε και για το χρονοδιάγραμμα των ε, τροπολογιών. <coughs> Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε να σας ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα για την συνεισφορά, συνεισφορά σας των ομιλητών, των σχεδόν ε, εισηγητών για τις ιδέες οι οποίες υπευλήθησαν και επίσης να ευχαριστήσω και το Κοινοβούλιο του Λουξεμβούργου για την επιστολή του. Η εντύπωσή μου είναι ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει όλους μας. Όλοι έχουμε εμπειρία από πρώτο χέρι για τα θέματα αυτά ως τακτικοί επιβάτες σε αεροπορικές εταιρείες. Νομίζω μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τις δικές μας εμπειρίες. Εγώ προσπάθησα παντά να διαφοροποιώ την δική μου προσωπική στάση βάσει της ε, προσωπικής μου εμπειρίας και ήθελα να ακούσω και την άποψη των άλλων. Έστειλα λοιπόν ερωτηματολόγια σε εταιρείε, σε αεροδρόμια, σε συνδικάτα κτλ. Και έχω προσπαθήσει να λάβω υπόψη όλες τις ιδέες και τις προτάσεις που μου έχουν υποβάλει και επίσης και τα πορίσματα συνδιασκέψεων και σεμιναρίων για τα θέματα αυτά. Χωρί ακόμα κάποια βεβαιότητα για τα ζητήματα αυτά φυσικά, αλλά προσπάθησα να μπω σε λεπτομεριακό επίπεδο στο βαθμό του δυνατού και συμφωνώ με τους συναδέλφους που λένε ότι οι υπηρεσίες εδάφους δεν είναι επαρκώς αποτελεσματικές λόγω κάποιων περιορισμών που εξακολουθούν να υπάρχουν. Και συμφωνώ και με αυτούς από εσά που έχουν υπογραμμίσει τη σημασία της ασφάλειας, μιλήσανε για την ποιότητα, για τα δικαιώματα των καταναλωτών. Εγώ βέβαια έχω περιορισμένες δυνατότητες επί τη βάση όλων των στοιχείων που έχω συλλέξει, έχω ένα περιορισμένο πλαίσιο να καταθέσω τροπολογίες που να απτώνται τις αρμοδιότητες της Επιτροπής μας. Και επομένως προσπάθησα να εστιάσω μονάχα στα θέματα που έχουν να κάνουν με αυτά που υπογραμμίσανε και οι σκιώδεις συζητητές. Παραδείγματος χάρη στη διαδικασία διαγωνισμών για να εξασφαλίσουμε για να πάροχο υπηρεσιών. Για να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη ποιότητα έχω κατατάξει σε τέσσερις ή πέντε κατηγορίες τις υπηρεσίες αυτές που μπορούν να την χάνουν ε, διαδικασίας ε, χωριστής η κάθε περιοχή αυτή. Αυτό θα μπορούσε να αυξήσει την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα με μια κατάτμιση των υπηρεσιών σε διάφορες <clears throat> υπηρεσίες οι οποίες θα υπέκυντο σε διαφορετικές διαδικασίες προσφορών. Μια δεύτερη ιδέα είναι αυτή των ελαχίστων προτύπων και εγώ συμφωνώ απόλυτα με αυτή την ιδέα και η ελπίδα μου είναι ότι οι πάροχοι θα μπορούσαν να ικανοποιήσουν αυτές τις ε, προδιαγραφές. Δεν έχω πολύ χρόνο και γι' αυτό τελικά σας ευχαριστώ για τις προτάσεις σας και την Κομισιόν για τα σχόλια που μας έδωσε και τις πληροφορίες. Είμαι προφανώς ανοιχτή για περαιτέρω συζήτηση και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να αποστάξουμε από όλες τις προτάσεις ένα σύνολο προτάσεων και θέσεων που θα είναι ικανοποιητικέ για όλους μας. Είμαστε απλώς μια γνωμοδοτική επιτροπή στο κάτω-κάτω. Εντάξει, λέω θα υπάρξει πολύ ενδιαφέρον για το θέμα αυτό και βασιζόμαστε σε εσά να παρουσιάσετε τη θέση μας στην Επιτροπή Μεταφορών. Προθεσμία τροπολογιών 18 Ιουνίου το μεσημέρι και στις 9 Ιουλίου θα συζητήσουμε αυτές τις τροπολογίες, θα ψηφίσουμε στις 10 ώστε να μπορέσει να έρθει στην Επιτροπή Μεταφορών το Σεπτέμβριο. Ευχαριστούμε κυρία Γκαλπέλτ και <clears throat> όλους τους σκιώδεις Προτού περάσουμε τώρα <clears throat> στη γνωμοδότηση του κυρίου Κουρέι Αντεκάμπου για τα ομόλογα σταθερότητα. θέλω να υπενθυμίσω αυτό που είπα προηγουμένως όταν δεν υπήρχαν πολλοί παρόντες. <clears throat> Αποφασίσαμε να ψηφίσουμε από κοινού στις 21 Ιουνίου δύο προτάσεις για πρώτη ανάγνωση. και όχι σήμερα προ, ε, προεβλέπετο να ψηφίσουμε και για την έκθεση του κυρίου Μπίελεν όπου έχουμε ήδη την αποδοχή από το Συμβούλιο των αποτελεσμάτων του τριγωνικού διαλόγου και θα έχουμε και την πρόταση προτυποποίησης από το Συμβούλιο. 21 Ιουνίου λοιπόν <clears throat> θα παρουσιάσουν οι δύο εισηγητές την θέση που προέκυψε από τη συνδιαλλαγή και θα πρέπει να κάνουμε την επίσημη έγκρισή τους. Και έτσι έχετε και δύο ακόμα εβδομάδες για να εξετάσετε αυτές τις προτάσεις. Χωρίς φυσικά να καθυστερήσουμε την Ολομέλεια, την έγκριση στην Ολομέλεια που ήταν το Σεπτέμβριο ούτως ή άλλως. Τον Ιούνιο θα ψηφίσουμε, έχουμε πολλά πράγματα να ψηφίσουμε. Θα σας πω τις ημερομηνίες στο τέλος, αλλά η γραμματεία θα σας ενημερώσει για όλα αυτά. Έχουμε κάνει πάρα πολλά τους τελευταίους μήνες και τώρα έχουν συγκεντρωθεί όλα αυτά τα στοιχεία τον Ιούνιο για τις ψηφοφορίες. Σίγουρα θα θέλετε να έχετε μία συνέχεια για το πακέτο προτάσεων και γνωμοδοτήσεων. Σχέδιο γνωμοδότηση για την Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή πρόκειται για μια έκθεση πρωτοβουλίας για το εφικτό της εισαγωγής ομολόγων σταθερότητος. Ο καθηγητής Κορία Δεκάμπους είναι ο εισηγητή μα και του δίνουμε χαρά το λόγο. Έχουμε την κυρία Βερχέιεν ω σκιώδη, τον κύριο Σμιτ δεν τον έχουμε, από ό,τι βλέπω. Η κυρία Ρούλα μπορεί να ξαναγυρίσει. Ο κύριος Φόξ θα παρουσιαστεί από κάποιον άλλο η θέση του. Καθηγητά Κουρέα Δεκάμπους, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να σας αναφέρω ποια είναι τα όρια του εγχειρήματο αυτού. Δεν πρόκειται για μία απόφαση για τα ομόλογα σταθερότητος, απλώς είναι μια γνωμοδότηση για το θέμα της, ε, του εφικτού της ε, δυνατότητας να υπάρξουν τέτοια ομόλογα. Η κυρία Φερχέιεν ζητάει το λόγο. Ναι, δεν έχετε μετάφραση. Χωρίς μικρόφωνο, κύριε Βερχέιεν. Ναι, ναι, ναι, λέει ο πρόεδρος. Δεν με ακούγατε, αλλά σας έχω εγγράψει στον κατάλογο των μιλτών γιατί είσαστε σκιώδης εισηγήτρια. Λοιπόν, λέει ο κύριος Κορέα Ντεκάμπους, όπως είναι γνωστό, η πολιτική μου ομάδα και εγώ ίδιος υποστηρίζουμε την εισαγωγή των ομολόγων σταθερότητας. Ένα από τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή οικονομία ήταν η πρόσβαση σε εύκολες πιστώσεις που οδήγησαν μετά την, το σπάσιμο της φούσκας το 2008 σε προβλήματα χρηματοδότησης. Ένα από τα μέτρα λοιπόν τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ξεπεραστεί το πρόβλημα αυτό είναι η ιδέα των ομολόγων σταθερότητας. Μπορούν να είναι ένα από τα κλειδιά που θα μπορέσουν να ξεκλειδώσουν τις δυσκολίες των κρατών μελών και ιδίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που βασίζονται στην ε, πίστοση, στις πιστώσεις τραπεζικές για να έχουν επενδύσεις και ανάπτυξη. Η Κομισιόν έχει κάνει μια εμπεριστατωμένη μελέτη η οποία έχει αντιμετωπίσει τα θέματα αυτά και υπάρχει και το έργο του Γερμανικού Ινστιτούτου Συμβούλων που, στο οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Όλι Ρεν πρόσφατα. Πιστεύουμε λοιπόν ότι πρέπει να συζητήσουμε όλες αυτές τις προτάσεις και να τις συγκρίνουμε και να δούμε κατά πόσο είναι πράγματι ε, εύστοχες οι επικρίσεις που αναφέρονται στα ομόλογα σταθερότητα. Πρέπει η Επιτροπή μας, η οποία είναι μια Επιτροπή που αφορά και τα θέματα των καταναλωτών, θα πρέπει να αντιμετωπίσει το θέμα της προστασίας των δικαιωμάτων των επενδυτών οι οποίοι, θα, οι οποίοι έχουν στα χέρια τους αυτή τη στιγμή ομόλογα χρέους του, των κρατών μελών. Αν τα νέα ομόλογα σταθερότητας έχουν υπέρτερο επίπεδο, είναι senior, έχουν προτεραιότητα δηλαδή σε σχέση με τα παλαιότερα ομόλογα, τι θα συμβεί για τους ομολογούς αυτούς. Επομένως πρέπει να αντιμετωπιστεί το θέμα μιας μεταβατικής ρύθμισης. Υποστηρίζουμε το να, είναι να έχουν προτεραιότητα τα ομόλογα σταθερότητα, αλλά θα πρέπει να καθοριστεί και η κατάσταση των τωρινών ομολογίουχων. Κάποια θέματα σε σχέση με την Πράσινη Βίβλο. Καταρχήν, η δυνατότητα τα κράτη-μέλη τα οποία δεν ε, πληρώνουν το χρέος τους να τεθούν υπό έλεγχο του, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν πρόκειται ε, μονάχα για αποθέματα τους σε χρυσό ή σε συνάλλαγμα, αλλά ακόμα και τα έσοδά τους από διάφορες υπηρεσίες θα πρέπει να τεθούν υπό έλεγχο. Αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι ένα θέμα το οποίο είναι ιδιαίτερα καυτό και ευαίσθητο σε χώρες οι οποίες βρίσκονται ήδη υπό κάποιο καθεστώς ε, εποπτείας. Πρέπει να λάβουμε επίψη στο τωρινό πολιτικό και οικονομικό πλαίσιο όπου ήδη για πολλές χώρες υπάρχει ε, μεγάλη πίεση και περιορισμή στην οικονομική δραστηριότητα για να υπόκειται κανείς στο μηχανισμό. Επίσης είναι απαραίτητο να υπάρχει και παράλληλη υποστήριξη για την επίλυση των προβλημάτων του προϋπολογισμού. Το επόμενο πρόβλημα έχει να κάνει με τη μετάβαση αυτού του, του συστήματος προς ένα σύστημα χρηματοδότησης από την αγορά. Πρέπει επίση να δούμε ποιο είναι το νομικό πλαίσιο για αυτά τα ομόλογα και ποιοι θα είναι αρμόδιοι σε περίπτωση διαφορών, για την επίλυση διαφορών, ώστε να μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχουν και μηχανισμοί υπεράσπιση των δικαιωμάτων των επενδυτών. Είμαι σίγουρο ότι η Κομισιόν θα είναι σε θέση να παρουσιάσει μια βιώσιμη και αποτελεσματική πρόταση και η συζήτησή μας θα συμβάλλει σε αυτό το αποτέλεσμα και ελπίζω ότι θα είναι δυνατόν να πείσουμε τις χώρες οι οποίες ακόμα είναι διστακτικές σε σχέση με αυτή την ιδέα. Και ελπίζω ότι η Επιτροπή μας θα έχει μια θετική γνώμη <clears throat> για το θέμα αυτό και θα συμβάλλει στην επίτευξη μια σωστή πρόταση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Για να επιβεβαιώσω, έχουμε την κυρία Βερχέν, σκιώδη για το ΕΛΚΟ, κύριος Μάντρης θα μιλήσει για τον κύριο Σμίτ, η κυρία Ρουρ είναι εδώ αυτή τη στιγμή. Έχω ένα γραπτό σχόλιο του κύριου Φόξ, το οποίο θα συνοψίσω για σας. Κύριε Βεχέιν πρώτα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον κύριο Κουρέιντ Κάμπς. Οι βασικές θέσεις της Κομισιόν στην Πράσινη Βίβλο <clears throat> είναι νομίζω μια βάση επί της οποίας μπορούμε να εργαστούμε. Δεν μπορούμε τώρα να πούμε ότι έχουν επιληθεί όλα τα θέματα, θα πρέπει <clears throat> να δούμε ποια θα είναι η πραγματική επίπτωση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις των ομολόγων σταθερότητος, ανεξάρτητα από το αν αυτό θα επιτύχει τη σταθεροποίηση των αγορών. Υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα τα οποία ε, εγείρονται σε σχέση με το εφικτό και το ρεαλιστικό των ομολόγων σταθερότητος και αν <clears throat> τελικά τα ομόλογα σταθερότητα θα πρέπει να τεθούν σε λειτουργία μονάχα μετά από το τέλος μιας μακράς διαδικασίας συμφωνιών και συντονισμού της οικονομικής πολιτικής. Σε σχέση με την πρόταση της Κομισιόν στην Πράσινη Βίβλο παραμένουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να επιληθούν ακόμα και να διευκρινιστούν και γι' αυτό νομίζω ότι η συζήτηση αυτή που θα λάβει η χώρα στην Οικονομική Επιτροπή θα είναι πάρα πολύ σημαντική και φυσικά θα προκύψουν και νέα ερωτήματα από αυτήν τη συζήτηση ώστε να ξεπεράσουμε αβεβαιότητες οι προσδοκίες οι οποίες θα είναι λανθασμένες. Έχουμε πολλές επιλογές από ό,τι αναφέρει η Κομισιόν στο εγγραφό της για τα ομόλογα σταθερότητα, οι οποίες είναι υποσυζήτηση, έχουν διαφορετικό χαρακτήρα και στην Πράσινη Βίβλο υπάρχει μια παρουσίαση και αξιολόγησή τους. Η πρώτη παραλλαγή είναι η πιο ριζοσπαστική, πιο ρηξικέλευτη και αυτή που περιέχει και περισσότερο κίνδυνο να ενώσουμε όλα τα ομόλογα των κρατών μελών και να έχουν ενιαία απόδοση, ενιαία δηλαδή επιτόκια. Δεν υπάρχει βεβαιότητα ότι αυτό θα μπορέσει να επιτευχθεί όμως, όπως λένε οι εμπειρογνώμονες, γιατί υπάρχει και το θέμα της ε, εμπιστοσύνης των αγορών. Η δεύτερη επιλογή αφορά μονάχα ένα τμήμα των ε, ομολόγων που θα τεθούν από κοινού και θα παραμείνει δυνατότητα τα κράτη-μέλη να έχουν δικά τους ομόλογα τα οποία θα έχουν διαφορετική απόδοση και διαφορετική ασφάλεια. Και εδώ χρειάζεται να υπάρξει περαιτέρω διευκρίνηση κάτω από ποιες προϋποθέσεις θα μπορούσε να είναι εφικτή μια τέτοια διαδικασία. Η τρίτη επιλογή, εδώ δεν χρειάζεται πολλή συζήτηση, γιατί ουσιαστικά είναι μια παράταση του τωρινού status quo και δεν οδηγεί σε μια ιδιαίτερη βελτίωση του καθεστώτος, όπου κάθε κράτος μέλος εκδίδει τα δικά του ομόλογα και αναλαμβάνει τη δική του ευθύνη. Και οι χρηματαγορές δεν έχουν δεν θα δώσουν ιδιαίτερη υποστήριξη σε ένα τέτοιο μοντέλο. Έχουμε τώρα σε όλες αυτές τις περιπτώσεις να αντιμετωπίσουμε τους κινδύνους πιστοτικής αφαιρεγγιότητος που πρέπει να καλυφθούν από τους φορολογούμενους και εδώ ή, όχι. Και εδώ θα πρέπει να μπορέσουμε να δούμε κατά πόσο θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση μιας συλλογικής ε, κάλυψης των απολειών αυτών. Το ερώτημα είναι αν μπορούμε να αντικαταστήσουμε τους μηχανισμούς της αγοράς από ένα μηχανισμό που θα είναι κατά ανάγκη γραφειοκρατικός. Επίσης είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε το κατά πόσον είναι απαραίτητες ε, αλλαγές των συνθηκών αν πρέπει να υπάρξουν παραδείγματος σε ορισμένα κράτη-μέλη αποφάσεις ε, εθνικών συνταγματικών δικαστηρίων που θα επιτρέψουν μια τέτοια ρύθμιση και την ανάληψη χρέους άλλων χωρών. Πιστεύω λοιπόν ότι με το σχέδιο του κυρίου Κουρέα Ντεκάμπους μπορούμε να προσθέσουμε και πρέπει να προσθέσουμε ορισμένα σημεία, να θέσουμε συγκεκριμένες ερωτήσεις. Από τη δική μας ε, πλευρά μέχρι τις 12 Ιουνίου θα έχουμε τις δικές μας προτάσεις να δώσουμε στον εισηγητή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ την κύριε Βερχέν. Ο κύριο Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη για τον κύριο Σμιτ επειδή έπρεπε να παρισταθεί στην ψηφοφορία της Επιτροπής ΕΚΟΝ. Θα διαβάσω ορισμένα σχόλια εκ μέρους του. Θα ήθελα να ευχαριστήσει την Αντώνιο για την έκθεσή του. Η έκθεση είναι πολύ ισορροπημένη και συμφωνεί ότι πρέπει να αξιολογηθούν όλες οι προτάσεις της ε, Πράσινης Βίβλου και του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων. Η προϋπόθεση για την κοινή έκδοση ομολόγων είναι ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν μειώσει τα τρέχοντα ελλείμματα και χρέη τους. Υπάρχει ανάγκη να υπάρχει ένα πλαίσιο δημοσιονομικής εξυγένσης. Ε, επίσης το ζήτημα του ηθικού κινδύνου θα πρέπει να αντιμετωπιστεί κατάλληλα ώστε το σύστημα να λειτουργήσει σωστά. Η Επιτροπή επίσης θα πρέπει να καθορίσει κριτήρια εισόδου και εξόδου βάσει σαφών προϋποθέσεων όπως δημοσιονομικής πειθαρχίας και αντιγωνιστικότητας. Τέλος, ο κύριος Σμιτ ε, ε, προέρχεται από χώρα που δεν ανήκει στην Ευρωζώνη. και η γνώμη εκεί για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αρκετά, η γνώμη του είναι αρκετά αρνητική αυτή τη στιγμή. Χρειάζεται λοιπόν να δημιουργήσουμε περισσότερη υποστήριξη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για το ευρώ. Θα ήθελε λοιπόν να τονίσει ότι είναι σημαντικό και αναγκαίο να γίνει δημοσία διαβούλευση για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της εισαγωγής ε, project bonds και θα πρέπει να υπάρξει έγκριση από το κοινό από τους πολίτες πριν εισαγαγούμε ομολογά σταθερότητα. Οι άνθρωποι φοβούνται για το μέλλον τους αυτή τη στιγμή. Ό,τι αποφασίζουμε στα όργανα εδώ στις Βρυξέλλες ε, πρέπει να κοινοποιούνται στους πολίτες ε, για τόσο σημαντικά ζητήματα όπως αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Να σας απαντήσω. Να ακούσουμε την απάντηση του κύριου Φόξ και μετά θα επανέλθουμε. Ο κ. Φόξ είναι εισηγητή και αυτός από χώρα που δεν συμμετέχει στην Ευρωζώνη. Αναγνωρίζει ωστόσο ότι η σταθερότητα της οικονομίας της Ευρωζώνης είναι σημαντική και για τις χώρες μέλη της Ευρωζώνης και για τις άλλες εκτός. Η ιδέα λοιπόν των ομολόγων σταθερότητας θα είναι σημαντική παρόλο που είναι επιφυλακτικός για ορισμένες πτυχές του θέματος. Και αυτά συμβαδίζουν και με άλλα σχόλια που έγιναν ήδη και οι επιφυλάξει του αναφέρονται στην πλήρη αντικατάσταση των ε, ε, δημοσίων ομολόγων με ευρωπαϊκά. Και υπάρχει και ηθικός κίνδυνος, θεωρίας. Μείωση δηλαδή τη δημοσιονομική πειθαρχία από πλευρά των χωρών μελών. Και απλώ να μετακινείται το χρέος χωρίς να αντιμετωπίζονται οι πραγματικές αιτίε που το έχουν προκαλέσει και ε, θεωρεί ότι τίθεται και θέματα εθνικής κυριαρχίας όπως είπαν και οι κύριοι Δεκάμπο και Βερχέρεν Ο κύριος Φόξ, ωστόσο, θα ήθελε να έλθει με την ευκαιρία αυτή και στις απόψεις πρέπει να εκφράσει η ΙΜΚΟ στη συζήτηση αυτή. Να υπενθυμίσει μεταξύ άλλων ότι εκτός από τα θέματα που τίθενται εδώ, ιδίως για την χρηματοδότηση μικρών και μεσών επιχειρήσεων, ότι υπάρχουν και άλλα εργαλεία για την χρηματοδότηση τέτοιων επιχειρήσεων που θα πρέπει να υποστηρίξουμε αλλά και η πρόσβαση στην ενιαία αγορά και η πρόσβαση στις δημόσιες προμήθειες και η εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες. Όλα αυτά είναι σημαντικά για τις μικρές και μεσές επιχειρήσεις. Και κυρίως η ατζέντα για την ανάπτυξη. Ο ρόλος της ενιαίας αγοράς μέσα στην ατζέντα για την ανάπτυξη που θεωρεί ότι πρέπει να ενταχθούν στο ευρωπαϊκό εξάμεινο μαζί και με μερικά άλλα εργαλεία πολιτικής που θεωρεί ότι είναι σημαντικά και ότι θα αποτελούν μια σημαντική συνεισφορά στη συζήτηση της Επιτροπής Προστασίας των Καταναλωτών και Ενιαίας Αγοράς. Θα στείλω αντίγραφο των σχολείων αυτών στον κύριο Κάμπος για να το λάβει υπόψη. Αυτή λοιπόν η απάντηση του κύριου Φόξ. Επανέρχομαι τώρα στην ιδιότητα του Προέδρου και Παρακαλώ να κάνουν σχόλια τα μέλη της Επιτροπής. Κύριε Βάιλερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ορισμένες από τις παρεμβάσεις με προσκαλούν να θυμίσω ότι η συζήτηση για το σύμφωνο σταθερότητος που διεξάγουμε τώρα μαζί με συναδέλφους άλλων επιτροπών γίνεται κυρίως διότι απέτυχε η αγορά. Δεν υπάρχει πλέον κοινωνικά ανεκτή α, κεφαλαία αγορά. Και εκπλήσωμαι που δεν τα απορρίπτει αυτά καταρχήν ο κύριος Φόξ, αλλά μάλλον σκέφτεται τι τροποποιήσεις μπορούμε να επιφέρουμε. Θα το σκεφτούμε και εμείς βέβαια αυτό. Το γεγονός όμως ότι όλοι όσοι είμαστε μέσα στην Ευρωζώνη και όσοι δεν είμαστε και αυτοί που θέλουν να μπουν και αυτοί που δεν θέλουν να μπουν ότι όλοι είμαστε συνυπεύθυνοι για τη σταθερότητα στην Ευρώπη, αυτό βεβαίω το βρίσκω σωστό. Σήμερα το πρωί στην τηλεόραση η καγκελάριό μου, α πω η, Γερμανία, η Γερμανίδα καγκελάριο καλύτερα, ότι στην επόμενη διάσκεψη κορυφή θα υποβάλει πρόταση για περισσότερη Ευρώπη σε ορισμένες πολιτικές, δημοσιονομική και οικονομική. Καλύτερο συντονισμό δηλαδή από ό,τι μέχρι τώρα. Αυτό βέβαια ηχεί ε, μεν θετικά, να δούμε όμως ποιες θα είναι οι προτάσεις. Δεύτερο, είμαι πεπισμένη ότι τα ομόλογα αυτά τελικώς έρχονται, θα έλθουν. Το ερώτημα είναι πώς. Και νομίζω ότι εδώ χρειαζόμαστε ακόμα πληροφόρηση και συζήτηση. Και γι' αυτό ρωτώ εάν η Επιτροπή Οικονομικών ως αρμόδια της προτίθεται να διεξαγάγει ακρόαση ή αν το έχει ήδη κάνει. Για να γνωρίζουμε και τι κάνουν οι άλλες παράλληλα εργαζόμενες επιτροπές, να μπορέσουμε να σταθμίσουμε τις διάφορες επιλογές και να δούμε τελώς πώς θα τα αποφασίσουμε. Αντώνιο, μήπως εσείς έχετε κάποια πληροφορία από την Επιτροπή ΕΚΟΝ. Άλλος κανείς. Ξέρω ότι είναι παρόν εκπρόσωπος της Κομισιόν. Θα ζητήσω μετά από τον εισηγητή να ολοκληρώσει και να απαντήσει και στις ερωτήσεις της κυρίας Βάιλερ. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους κύριε Πρόεδρε που αυτούς που έχουν συμβάλει στη συζήτηση για το θέμα αυτό ιδίως την κυρία Φερχάιεν από το ΕΛΚ η οποία έθιξε το βασικό πρόβλημα του νομικού πλαισίου και το κατά πόσο αυτές οι παραλλαγές οι οποίες προτείνονται θα είναι συνταγματικά βιώσιμες. Το θέμα όμως του συνταγματικού πλαισίου τέθη ήδη το 2010 όταν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μπήκε στη δευτερογενή αγορά ομολόγων. Υπήρχαν προβλήματα, αλλά έγινε αυτό παρόλα αυτά. Όλα αυτά λοιπόν τα νομικά προβλήματα θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε ε, μέσα στο πλαίσιο μιας συνεχούς εξέλιξης των θέσεών μας. Κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα τουλάχιστον, αλλάζει η κατάσταση και αλλάζει η αντιμετώπιση. Επομένως, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η πρόταση του Γερμανικού Συμβουλίου ε, Οικονομικών Συμβούλων. Δεν είχα το χρόνο να διεξέλθω αυτή την πρόταση, αλλά σίγουρα θα χρειαστεί να επανέλθουμε στο θέμα αυτό στο μέλλον. Επομένως, σε σχέση με το νομικό πλαίσιο, θα πρέπει πραγματικά να το επεξεργαστούμε. Η παραλλαγή 3 που παρουσίασε η κυρία Φερχάιεν είναι κατά πάσα πιθανότητα η παραλλαγή αυτή η οποία δεν θίγει καθόλου την τωρινή συνταγματική τάξη αλλά είναι και η λιγότερο ε, αποδεκτή γιατί οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα δεχόντουσαν πολύ εύκολα να παραδώσουν την οικονομική τους κυριαρχία σε σχέση με τα έσοδά τους ή με το χρυσό στην κεντρική τους τράπεζα. Δεν πρέπει όμως να απορρίψουμε ακόμα καμία δυνατότητα, καμία παραλλαγή, γιατί ακόμα βρισκόμαστε σε μια διαδικασία μάθησης. Για τον κύριο Μάντερς. Θέλω να υπογραμμίσω κάτι από αυτά που είπε. Το βασικό θέμα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε είναι η εδραίωση των εθνικών προϋπολογισμών. Αυτό είναι απαράγραπτο. Επομένω, η συνένεση που δημιουργήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τι υποχρεώσει αυτέ των κρατών μελών και το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο είναι πράγματα τα οποία δεν θέτω σε συζήτηση. Είναι αδιαμφισβήτητα. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει το κατάλληλο πλαίσιο ώστε όλοι να κινηθούμε προς την κατεύθυνση της παγιοποίησης των δημοσιονομικών μας η πολιτική συζήτηση είναι εν εξέλιξη. Κάθε μέρα γίνονται συζητήσεις για τα θέματα αυτά. Και εγώ είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένο και θετικά εκπλήσωμαι για αυτά που είπε ο κύριος Φόξ για την έκθεση αυτή. Αν γυρίσουμε 2,5-3 χρόνια πριν, όταν ρίφθη για πρώτη φορά η ιδέα αυτή, υπήρξαν πάρα πολλοί έντονες αντιδράσεις από τους πολιτικούς ηγέτες και από τον πρόεδρο της Κομισιόν ακόμα που ήταν διαρρήδιν αντίθετη με τα ευρωομόλογα ή τα ε, ομόλογα σταθερότητας που λέγονται πια ευρωομόλογα και απλώς είχαν προτείνει σαν εναλλακτική λύση τα λεγόμενα ομόλογα έργου, τα project bonds. Τώρα όμως μετά από όλα αυτά, μετά από δύο χρόνια, έχει η Κομισιόν μια πρακτική πρόταση επί της οποίας μπορούμε να εργαστούμε. Έχει υπάρξει λοιπόν μια σημαντική πρόοδος και εξέλιξη απόψεων και ξέρουμε όλοι ότι η επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε <clears throat> για τη σταθεροποίηση του κρατικού χρέους είναι απαραίτητη για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε την ύφεση και να χρηματοδοτήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αυτό δεν αφορά μονάχα τις χώρες οι οποίες <clears throat> είναι ασθενείς τώρα αλλά και αυτές οι οποίες έχουν εμπορικό πλεόνασμα και παρόλα αυτά αρχίζουν τώρα να αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Τέλος, δεν θέλω να παραλείψω να αναφέρω σχετικά και την έννοια που αναφέρθηκε προηγουμένως, όχι από την κυρία Στήλερ, συγγνώμη, την κυρία Βάιλερ, συγγνώμη, συγγνώμη, μας τόνισε ότι κάθε μέρα υπάρχουν νέες ανακοινώσεις στα μέσα ενημέρωσης για τα θέματα αυτά. Και περιμένουμε όλοι προτάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν πρέπει να κάνουμε μελλοντολογικές αναλύσεις, αλλά πιστεύω ότι επίκυνται αυτές οι προτάσεις, ίσως όχι ως ε, ομόλογα σταθερότητος, αλλά ως ταμείο, κοινό ταμείο απόσβεσης χρέους ή με κάποιο άλλο με κάποια άλλη διατύπωση, ακολουθώντας κάποιες από τις εναλλακτικέ προτάσεις του Γερμανικού Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων. Γίνεται λοιπόν ήδη η κίνηση προς την κατεύθυνση αυτή, γιατί είναι θέμα ζωής και θανάτου σε δημοσιονομικό επίπεδο και οικονομικής επιβίωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Good. Um, thank Ευχαριστούμε πολύ. Απάντησε την ερώτησή σας, είστε ικανοποιημένοι. Ναι, αλλά τι γίνεται με την ΕΚΟΝ. Ε, Από ό,τι γνωρίζω, δεν έχει ακόμα επίσημη θέση η Οικονομική Επιτροπή για τα θέματα αυτά. Δεν νομίζω ότι έχει συζητηθεί επαρκώς το θέμα αυτό. Έχουμε πολλέ ερωτήσει, πολλά θέματα να εξετάσουμε, αλλά δεν έχουμε ακόμα οριστικέ απαντήσει. Ευχαριστώ. Ωραία, ευχαριστούμε. Απλά ήθελα να βεβαιωθώ, επειδή έχω και τις σημειώσεις, δεν έχω τη σημείωση του κ. Φόξ μπροστά μου, υπενιστεί ότι συμφωνεί με την πρόταση, λέει στην πραγματικότητα ότι κάποια ανάλυση των πιθανών πλέον εκτιμάτων τη εισαγωγή των ομολόγων σταθερότητα μεταξύ άλλων προτάσεων ίσω αξίζει κάποια σκέψη είναι κάτι νέο αυτό. Ήθελα να είμαι βέβαιος ότι προσφέρουμε σωστά τις προτάσεις του κ. Φόξ. Ευχαριστώ λοιπόν όλους σας ε, το χρονοδιάγραμμα. Τώρα προθεσμία για τις τροπολογίες είναι η 12η Ιουνίου για την εκτίση του κυρίου Ντεκάμπος ε, στις 12 το μεσημέρι. 9 Ιουλίου θα εξεταστούν οι τροπολογίε και 10 του μήνα θα ψηφιστούν. Θα είναι λοιπόν ε, οι μέρε στι οποίε θα είμαστε πολύ απασχολημένοι, γιατί έχουμε πολλέ γνωμοδοτήσει πριν από τι καλοκαιρινέ και το χρονοδιάγραμμα για την ΕΚΟΝ είναι το Σεπτέμβριο. Ωραία, λοιπόν, περνάμε τώρα σε μια εξαιρετική προσκεκλημένη, ένα ιδιαίτερο σημείο στη σημερινή σε διάταξη. Πάντα χαίρομαι όταν καλωσορίζω την κυρία Ζακλίν Μίνο, διευθύντρια με για θέματα καταναλωτών. Όπως γνωρίζετε όλοι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επισκέπτεται τακτικά την Επιτροπή μας και την ευχαριστούμε που είναι πάντα τόσο πρόθυμη να μας ε, μοιραστεί μαζί μας πληροφορίες ε, ώστε να μας βοηθήσει στο έργο μας. Όπως θα γνωρίζετε όλοι, πιστεύω, παρακολουθούμε στενά από την αρχή και τώρα βρισκόμαστε στην 7η έκδοση του πίνακα αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές. Πρόκειται για κάτι πλέον που έχει καθιερωθεί και το οποίο ενημερώνεται κάθε χρόνο όσο ονομάζεται «Οι καταναλωτέ στα σπίτια του στην ενιαία αγορά, παρακολούθηση της ενοποίηση τη ενιαία αγορά και των συνθήκων». Δεν είμαι βέβαιο κατά πόσο έχετε κάποιες διαφάνειες. Α, ετοιμάζουμε φωτοτυπίες. Φοβερή τεχνολογία σε αυτό το κτίριο. Ε, θα χρειαστεί να πληρώσουμε για τις φωτοτυπίες. Ε, θα μπορούμε να έχουμε λοιπόν τις φωτοτυπίες αυτές να τα επιτέγματα της τεχνολογίας. Ε, ξεκινάμε λοιπόν με ένα ελαφρύ μειονέκτημα, δεν έχουμε τα αντίγραφα, αλλά μπορούμε να προχωρήσουμε και στη συνέχεια μπορείτε να κάνετε σχόλια καθώς θα προχωρούμε. Οπότε φροντίστε να τραβήξετε την προσοχή μου. Ζακλίν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ που μας ε, καλέσατε να παρουσιάσουμε αυτό τον 7ο πίνακα αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές στην Επιτροπή σας. Καθώς ε, συζητάμε αυτή τη στιγμή, οι φωτοτυπίες ε, του αρχείου μου, του PowerPoint, ετοιμάζονται. Θα είναι λίγο δύσκολο να ακολουθήσετε χωρίς τις φωτοτυπίες, αλλά τα περισσότερα από όσα θα πω αντιστοιχούν ε, σε πίνακες που υπάρχουν μέσα στο έγγραφο. Το έχετε αυτό το έγγραφο μπροστά σας? Όχι. Λοιπόν, θα κάνω ό,τι μπορώ καλύτερο. Όπως πιστεύω γνωρίζετε όλοι σας, ο πίνακας αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές είναι ένα εργαλείο παρακολούθησης της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και των αγορών γενικότερα από την άποψη των καταναλωτών. Για εμάς ε, αποτελεί ένα εργαλείο κλειδί διότι μας παρέχει αποδεκτικά στοιχεία. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι κάθε πολιτική θα πρέπει να βασίζεται σε στοιχεία και αποδεκτικά στοιχεία. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τα αποτελέσματα για τους καταναλωτές που έχουν οι κανονισμοί της εσωτερικής αγοράς. Αυτό που κάνουμε λοιπόν είναι ότι παίρνουμε τη θέση των καταναλωτών στην εσωτερική αγορά και ελπίζουμε αυτό να τροφοδοτεί όλα τα στοιχεία που συλλέγουμε τις ε, συζητήσεις πολιτική Ο πίνακα. δημοσιεύεται δύο φορές το χρόνο, μία φορά το φθινόπωρο όπου εξετάζονται 50 διαφορετικές ε, αγορές καταναλωτών, διαφορετικές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών. Τις εξετάζουμε από άψη εμπιστοσύνη, συγκρισιμότητα, συνολική ικανοποίηση, ώστε να εντοπίσουμε τους τομείς με την καλύτερη απόδοση και τους τομείς με λυπή απόδοση που ενδεχομένως ε, χρήζουν περισσότερης προσοχής ε, από όσους χαράσουν πολιτική. Αυτός ο πίνακας αποτελεσμάτων, που είναι ο έρηνος πίνακας αποτελεσμάτων, εξετάζει κάποιους διαφορετικούς τομείς ενδιαφέροντος. Εξετάζουμε συγκεκριμένα δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι αναλύουμε τι ε, συνθήκε για του καταναλωτέ, στα κράτη-μέλη, το περιβάλλον για του καταναλωτέ, το περιβάλλον μέσα στο οποίο οι καταναλωτέ ε, δραστηριοποιούνται καθημερινά. Πόση εμπιστοσύνη έχουν στι δημόσιε αρχέ, πώς, ε, ποια είναι η άποψή του για του λιανοπολιτές, αν θεωρούν ότι τα προϊόντα που βρίσκουν στα σούπερ μάρκετ του είναι ασφαλή. Αυτό είναι ένα τομέα που εξετάζουμε και θα επανέλθω σε αυτόν, ο δεύτερο τομέα είναι το διοσυνοριακό εμπόριο και το ηλεκτρονικό εμπόριο. Χρησιμοποιούν οι Ευρωπαίοι πράγματι την ενιαία αγορά ώστε να αγοράζουν προϊόντα και υπηρεσίες από χώρες ε, εκτός της χώρας ε, διαμονής τους. Και αυτό μας επιτρέπει να αξιολογήσουμε την ενοποίηση της εσωτερικής ε, αγοράς στην Ευρώπη και ειδικότερα της ηλεκτρονικής αγοράς. Πρώτα απ' όλα λοιπόν οι συνθήκες για τους καταναλωτές τι άποψη έχουν οι καταναλωτές όσον αφορά το περιβάλλον μέσα στο οποίο πρέπει να λαμβάνουν καθημερινά αποφάσεις για την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών. Ε, εδώ δημιουργούμε ένα ευρετηρίο συνθήκων των καταναλωτών με σκοπό να έχουμε μέσα στο χρόνο ένα σύνολο στοιχείων το οποίο φυσικά εμείς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αλλά το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από ε, Όσου χαράσουν πολιτική σε εθνικό επίπεδο και άλλου ενδιαφερομένους για τον καθορισμό των επιπτώσεων των πολιτικών στην ευημερία των πολιτών. Έχουμε τώρα ένα τριετές ε, χρονικό διάστημα, οπότε μπορούμε να παρατηρούμε, να παρακολουθούμε την εξέλιξη των μεσονόρων, των συνθηκών στα διάφορα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη μπορούν να ε, θέτουν ε, ως benchmark τους καλύτερους οι χώρες που θεωρούνται συγκρίσιμες από ψυχιογραφική και οικονομικής ανάπτυξης και όσον αφορά και το μέγεθος της αγοράς. Βασίζουμε το ευρετήριο αυτό σε έρευνες που πραγματοποιούμε μεταξύ καταναλωτών και ελληνοπολιτών. Αποτελείται συνολικά από 12 στοιχεία τα οποία σχετίζονται με την ποιότητα του κανονισμού, όσο και με την επιβολή. Αν είχατε τώρα τη διαφάνεια μπροστά σας θα μπορούσατε να δείτε αυτά τα 12 στοιχεία, θα σας τα περιγράψω γρήγορα. Εξετάζουμε την ικανοποίηση με τα υπάρχοντα μέτρα προστασίας των καταναλωτών, την ύπαρξη παραπλανητικών διαφημίσεων ή προσφορών και τις ε, απάτες σε πλαίσια προσφορών και διαφήμισης όσον αφορά την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Μιλάμε για την εμπιστοσύνη τους στις δημόσιες αρχές Στου ε, πολιτέ και παρόχου υπηρεσιών, δηλαδή στου λιανοπολιτέ, κατά πόσο πιστεύουν ότι γενικότερα οι επιχειρήσει ανταποκρίνονται στι ανησυχίε και ανάγκε των καταναλωτών. Εξετάζουμε επίση την εμπιστοσύνη του, στι οργανώσει καταναλωτών. Ω τρίτο στοιχείο εξετάζουμε τι ε, διαμαρτυρίε. Θεωρούν δηλαδή ότι ε, αξίζει τον κόπο να υποβάλουν παράπονα οι καταναλωτές. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. αν αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι ένα πρόβλημα απλά να σηκώνουν τους ώμους και το αποδέχονται ως κομμάτι της καθημερινότητας. Ε, αυτό φυσικά δεν τους ενδυναμώνει ιδιαίτερα. Ε, εξετάζουμε την ικανοποίηση από την εξέταση παραπώνων, την επίλυση διαφορών και τέλος την ασφάλεια των προϊόντων. Τα δεδομένα αυτά σχετίζονται με το 2011. Τι συνέβη λοιπόν σε αυτό το έτος. Στο σύνολο έχουμε κάποια καλά νέα. Για έξι από αυτά τα δώδεκα στοιχεία παρατηρήθηκε θετική πρόοδος. Τα πράγματα έχουν βελτιωθεί. Έξι από αυτούς τους δείκτες λοιπόν έχουν ανέλθει. Ε, τρεις παρέμειναν σε ίδια επίπεδα και τρεις υποβαθμίστηκαν. Μόνο σε τρία στοιχεία λοιπόν παρατηρήθηκε η υποβάθμιση των συνθήκων των καταναλωτών. Δύο από αυτούς τους ε, τρεις δείκτες που πήγαν στο κόκκινο σχετίζονται με την ασφάλεια των προϊόντων που ανησυχεί τόσο τους καταναλωτές όσο και τους λιανοπολίτες οι οποίοι έχουν την αίσθηση ότι η ασφάλεια των προϊόντων έχει υποβαθμιστεί κατά το τελευταίο έτος. Κοιτώντα το συνολικό, το όλο ευρετήριο, στο σύνολο υπάρχουν κάποια καλά νέα. Το ευρετήριο καταδεικνύει μια ελαφριά βελτίωση των συνθήκων για τους καταναλωτές στα περισσότερα κράτη-μέλη. Στα 19 από τα 27 κράτη-μέλη τα πράγματα έχουν βελτιωθεί από απόψη όσον αφορά την αντίληψη των ε, καταναλωτών και των γιανοπολιτών σε σχέση με το 2010. Πρέπει να πω ότι έτσι συνεχίζεται η αναβάθμιση μετά από μια τεράστια πτώση το 2009. Το 2009 παρατηρήθηκε μια τεράστια υποβαθμίση όλων αυτών των δικτών. Όλα πήγαν στο κόκκινο. Πέρυσι παρατηρήθηκε, σημειώθηκε κάποια πρόοδος, κάποια επαναφορά της εμπιστοσύνης, η οποία συνεχίζεται φέτος, με λίγο βέβαια πιο αργούς ρυθμούς. Τα κράτη-μέλη στα οποία παρατηρήθηκαν οι σημαντικότερες βελτιώσεις ε, βελτιώσεις της τάξης του 6% ήταν η Βουλγαρία, το Βέλγιο, η Γαλλία και η Δανία. Σε αυτές τις χώρες δηλαδή σημειώθηκαν σημαντικά βελτιωμένες ε, συνθήκες. Φυσικά εξακολουθούμε να, εξακολουθούν να σημαίνονται δύσκολες δημοσιονομικές και οικονομικές συνθήκες με αρνητικές επιπτώσεις ορισμένα κράτη-μέλης Τέσσερα κράτη-μέλη, Ιταλία, Σλοβενία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία σημειώθηκε η υποβάθμιση της ποιότητας του περιβάλλοντος για τους καταναλωτές και σε τέσσερις άλλες χώρες τα πράγματα δεν άλλαξαν ιδιαίτερα Πολωνία, Κύπρος, Πορτογαλία και Σλοβακία. Αυτή είναι λοιπόν η πρόοδος για το 2011. με απόλυτου όρου. Πρέπει να διασαφηνίσουμε ότι ο σκοπό του πίνακα αποτελεσμάτων δεν είναι να στιγματίσει χώρες. Α, η τεχνολογία κάνει την εμφάνισή τη. Ευχαριστούμε. Δεν έχει λοιπόν σκοπό ο αποτελεσμάτων να στιγματίσει κάποιες χώρες, αλλά προσπαθούμε να εντοπίσουμε τις βέλτιστες πρακτικές, ώστε να μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι χώρες που φαίνεται να τα πηγαίνουν καλά, τι μπορούν να μας διδάξουν. Οι καλύτερε συνθήκε, όπω φαίνεται, βρίσκονται στο Λουξεμβούργο, το Ενωμένο Βασίλειο, τη Δανία, την Αυστρία, την Ιρλανδία, τη Φιλανδία, τι κατοχώρε, το Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Σουηδία με αυτή τη σειρά. Εάν προσέξατε αυτή τη λίστα θα παρατηρήσετε ότι μιλάμε για χώρε της Βορειοδυτική Ευρώπη και ότι πρόκειται για τα παλιότερα κράτη-μέλη. Αυτό που προκύπτει λοιπόν πολύ σαφώ από αυτό το πίνακα αποτελεσμάτων είναι ότι έχουμε ένα διαχωρισμό βορειοδυτικών και νοτιοανατολικών χωρών. Οι καλύτερες συνθήκες ε, παρατηρούνται συστηματικά στο βόρειο και δυτικό κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι πιο υποβεθμισμένες συνθήκες στο νότιο και ανατολικό. Αθέμητες εμπορικές πρακτικές για αυτό το θέμα Ρωτάμε κατά πόσο υπάρχουν ως επιτοπλίστων αθέμητες εμπορικές πρακτικές. Θέλουμε να δούμε κατά πόσο οι καταναλωτές και οι λιανόπολιτες θεωρούν ότι οι αγορές ε, αποδίδουν ε, όπως θα πρέπει κατά πόσο έχουν αποκλειστεί οι αθέμητες πρακτικές από την αγορά είναι κρίσιμη σημασία φυσικά τόσο για τους καταναλωτές να προστατεύονται από αθέμητες εμπορικές πρακτικές αλλά είναι και σημαντικό για τις ε, ε, καλής φήμης επιχειρήσεις ε, το να μην έχουν ανταγωνιστές που εξαπατούν ή παραπλανούν τους καταναλωτές θα πρέπει αυτοί να εξελιχθούν από την αγορά μας ανησυχεί λοιπόν ότι το 2011 υπήρξε αντιληπτή αύξηση των αθέμητων περιπτώσεων ε, των περιπτώσεων αθέμητου εμπορίου τόσο μεταξύ καταναλωτών όσο και μεταξύ λιανοπολιτών. Ρωτήθηκαν λοιπόν καταναλωτέ κατά πόσο έχουν έρθει σε επαφή με παραπλανητικέ ή απατηλέ διαφημίσει ή διαφημίσει που δεν έχουν ζητηθεί και οι λιανοπολιτέ ρωτήθηκαν κατά πόσο γνώριζαν ανταγωνιστέ οι οποίοι εξασκούν πρακτικές παραπλάνησης, παραπλανητικής διαφήμισης ή άλλης εμπορικής επικοινωνίας και τα αποτελέσματα δείχνουν αύξηση και για τις δύο πλευρές. Και οι δύο πλευρές αντιλαμβάνονται, παρατηρούν αύξηση αυτών των αθέμπτων πρακτικών. Αυτό φυσικά αποτελεί για εμάς λόγο ανησυχίας και καταδεικνύει την ανάγκη να συνεχίσουμε να επιμείνουμε στη βελτίωση της επιβολής ε, τόσο από το δημόσιο τομέα όσο και, μηχανισμούς, όσο και των μηχανισμών προσφυγής. Εξετάζουμε επίση την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Παρά το γεγονό ότι οι άνθρωποι έχουν έρθει σε επαφή με περισσότερε παραπλανητικέ πρακτικέ, η εμπιστοσύνη των καταναλωτών αυξάνεται. Παρότι ορισμένα πράγματα δεν πάνε καλά, η συνολική ικανοποίηση όσον αφορά τα μέτρα προστασία των καταναλωτών και τα επίπεδα εμπιστοσύνη στους διάφορους ε, ε, φορείς, δημόσιες αρχές, τους λιανοπολιτές, τους ίδιους και τους οργανισμούς καταναλωτών έχει σημειώσει σταθερή βελτίωση από το 2008 και εξακολουθεί να βελτιώνεται η εμπιστοσύνη των οργανισμών για τους οργανισμούς καταναλωτών και τις δημόσιες αρχές σημειώνει αύξηση κατά 8 εκατοστιαίες μονάδες. Μάλιστα, η εμπιστοσύνη προς τους παρόχους υπηρεσιών και τους πολιτές προϊόντων έχει αυξηθεί κατά 6%. Αυτό σημαίνει αύξηση λοιπόν της συνολικής ικανοποίηση για τις ε, καταναλωτικές αγορές και τα μέτρα προστασίας των καταναλωτών. Δεν δουλεύει, δεν δουλεύει το μαραφέτη αυτό. Μάλλον δεν φαίνεται η εικόνα.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 βρούμε σύντομα, ελπίζω, μια λύση για αυτό το ζήτημα. Τώρα, τώρα μιλούσα για την αυξή τη εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Ωστόσο, η συνολική ικανοποίηση κρύβει τεράστιε διαφορέ μεταξύ των κρατών μελών. Στη διαφάνεια που κανονικά θα βλέπατε τώρα, θα βλέπατε μια μείωση το 8% των καταναλωτών στην Αυστρία και στη Δανία έχουν εμπιστοσύνη στις δημοσίες αρχές, στους λιανοπολιτές, τους οργανισμούς προστασίας των καταναλωτών στην άλλη άκρη. Έχουμε χώρες στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, Ελλάδα, Βουλγαρία, Λιθουανία και Σλοβακία όπου τα επίπεδα εμπιστοσύνης έπεσαν ε, κατά 30%, στο 30%. Λιγότεροι από ένα στους τρεις καταναλωτές έχουν εμπιστοσύνη στο ότι θα υπερασπίσει κάποιος σωστά τα δικαιώματά τους. Κοιτώντας τον πίνακα αποτελεσμάτων που υπάρχει διαθέσιμος online, υπάρχουν δελτία για κάθε κράτος μέλος. Μπορείτε λοιπόν να δείτε και για το δικό σας κράτος μέλος ποιες είναι οι επιδόσεις ε, για καθένα από αυτά τα μέτρα. Περνώντας τώρα στην ασφάλεια των προϊόντων, είχα πει ότι αυτό ήταν ο ένας δείκτης που βρέθηκε στο κόκκινο. Και εδώ είναι ενδιαφέρον. Παρατηρούμε ότι συμπίπτουν οι απόψεις των καταναλωτών και των λιανών πολιτών. Και οι δύο θεωρούν ε, ότι υποβαθμίστηκε η ασφάλεια των προϊόντων εντός της ενιαίας αγοράς παρότι οι καταναλωτές είναι λίγο πιο απεσιόδοξοι από τους λιανοπολιτές. Οι καταναλωτές ανησυχούν περισσότερο. Σχεδόν οι μισοί καταναλωτές στη Ρουμανία και στην Ελλάδα θεωρούν ότι μεγάλος αριθμός προϊόντων δεν είναι ασφαλής πραγματικά δεν εμπιστεύονται τα αγαθά, τα προϊόντα στις αγορές τους ε, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό είναι 10% μόνο στη Φιλανδία, στις κατοχώρες και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πιστεύω ότι αυτό θα πρέπει να, να αντιμετωπιστεί με τους κανόνες παρακολούθησης της αγοράς αλλά και με την κοινή χρήση εμπειρογνώμοσύνης σωστών πρακτικών και εμπειρίας μεταξύ των κρατών μελών. Τι κάνουν σωστά οι αρχές στη Φιλανδία και στις κατοχώρες και τι πρέπει από μένα να κάνουν οι αρχές στη Ρουμανία και στην Ελλάδα. Φυσικά υπάρχει το ζήτημα των πόρων που αφιερώνονται στην ασφάλεια των προϊόντων, στην προστασία των καταναλωτών γενικότερα. Και πάλι στο έγγραφο αυτό θα βρείτε λεπτομερή στοιχεία για τον προ... κομμάτι του προπολογισμού, τον προπολογισμό που αφιερώνει κάθε κράτο μέλο σε αυτόν τον τομέα υπάρχει μια κλιμακωτή παρουσίαση βάσει και του μεγέθου τη αγορά. Συνεπώ, υπάρχει μια απευθεία σύγκριση μεταξύ κρατών μελών. Πιστεύω ότι θα πρέπει προσεκτικά να χρησιμοποιούμε αυτέ τι πληροφορίε. Είναι πολύ δύσκολο για τα κράτη-μέλη να αξιολογήσουν πόσο ακριβώ ξοδεύουν για την παρακολούθηση τη αγορά, για την επιτήρηση τη αγορά. Συχνά πρόκειται για τοπική ή περιφερειακή ευθύνη. Είναι λοιπόν δύσκολη συλλογή δεδομένων. Θα θυμάστε πιθανώς ε, πριν από 18 μήνες σας παρουσιάσαμε μία έρευνα για την ικανότητα των καταναλωτών που κατέδειξε ανησυχία όσον αφορά τις ικανότητες των καταναλωτών να κατανοήσουν τις πληροφορίες σε ετικέτες, να αναγνωρίσουν διάφορα σήματα. Είχαμε σχετικές ερωτήσεις στον πίνακα αποτελεσμάτων και δυστυχώς δεν μας καθησυχάζουν ιδιαίτερα. Οι καταναλωτέ νομίζουν ότι γνωρίζουν τα δικαιώματά του, αλλά όταν του ρωτάμε ουσιαστικά να απαντήσουν σε συγκεκριμένε ερωτήσει όσον αφορά τα δικαιώματα επιστροφή ενό προϊόντο, το κατά πόσο έχουν το δικαίωμα επανόρθωση, αντικατάσταση ενό προϊόντο ή ε, επισκευή ενό προϊόντο που έχει χαλάσει, μόνο το 30% των ερωτηθέντων κατάφεραν να απαντήσουν και τι τρει ερωτήσει, σωστά. Παρότι λοιπόν οι άνθρωποι θεωρούν ότι γνωρίζουν τα δικαιώματά τους, στην πραγματικότητα πολύ συχνά κάνουν λάθος. Το 12% σχεδόν ίδιο αριθμός δεν μπορούσε να απαντήσει σωστά σε καμία από τις ερωτήσεις. Υπάρχουν λοιπόν πολλές ε, διαφορετικές απόψεις ε, όσον αφορά το τι είναι δικαιώματα καταναλωτών. Επίσης οι λιανοπολιτές ε, ισχυριζόνται ότι σέβονται τα δικαιώματα των καταναλωτών. Όταν τους ρωτάμε αν εσείς ως ε, λιανοπολιτές σέβεστε τους ε, κανόνες προστασίας των καταναλωτών, το 95% λέει ναι, φυσικά αυτό δεν μας εκπλήσει. Αλλά όταν τους ρωτάμε λεπτομερείς ερωτήσεις όσον αφορά τις νομικές τους υποχρεώσεις, οι απαντήσεις τους είναι λανθασμένες. Για παράδειγμα, μόνο ένας από τους τρεις λιανοπολιτές γνώριζε πραγματικά το πόσο μεγάλη είναι η περίοδος ψύχρανσης, το cooling off περίοδο και μόνο ένας στου πέντε απλών λιανοπολιτών γνώριζαν την περίοδο εγγύησης κατά την οποία οι καταναλωτέ έχουν το δικαίωμα να επιστρέψουν ένα ελαττωματικό προϊόν. Και σε αυτή την περίπτωση λοιπόν πιστεύω ότι θα πρέπει να προσέξουμε και να μην θεωρήσουμε δεδομένο ότι οι επιχειρήσεις και οι λιανοπολιτές έχουν τις, γνωρίζουν και κατανοούν καλά τους κανόνες που εφαρμόζονται στην αγορά όπως ε, ισχυρίζονται. Λοιπόν, για όσους σας βλάβατε τώρα αντίγραφα των διαφανειών, έχω φτάσει στη διαφάνεια 11 που βρίσκεται στην κορυφή της σελίδας 6. Ε, Η επόμενη διαφάνεια, λοιπόν, διαφάνεια 12, ασχολείται με προβλήματα και παράπονα. Ένα ενδυναμωμένο καταναλωτέ και όλοι προσπαθούμε να ενδυναμώσουμε του καταναλωτέ, όχι μόνο γνωρίζει τα δικαιώματά του και όπω μόλι είπα δεν τα γνωρίζει απαραίτητα. Επίση δεν φοβάται να διαμαρτυρηθεί σε περίπτωση μη τήρηση σεβασμού αυτού των δικαιωμάτων του και δεν διστάζει να ζητήσει ε, να ε, προσφύγει ώστε να ζητήσει επανόρθωση η προθυμία των καταναλωτών να διαμαρτυρηθούν έχει σημειώσει σταθερή αύξηση μέσα στα χρόνια. Θα παρατηρήσετε στο γράφημα στη σελίδα 12 της διαφάνειας σιγά σιγά οι καταναλωτές είναι όλο και πιο ικανοποιημένοι με τον τρόπο αντιμετώπισης των παραπώνων τους από τους λιανοπολιτές αυτό σημαίνει ότι ανταποκρίνονται καλύτερα πλέον οι λιανοπολιτές, ότι ε, επιθυμούν να διατηρούν την εμπιστοσύνη, των, ε, την πίστη των καταναλωτών, των πελατών τους και χειρίζουν, προσπαθούν να χειρίζονται τα παράπονα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ένα πράγμα που εξακολουθεί να μας ανησυχεί ωστόσο είναι ότι εάν ένας καταναλωτής ε, δεν καταφέρει να ξεπεράσει το πρώτο εμπόδιο, δηλαδή δεν τον ικανοποιήσει ο λιανοπολιτής, θεωρούν ότι δεν τα κατάφεραν και τα παρατούν. Σταματούν λοιπόν εκεί. Αυτό σημαίνει ότι πολλά προβλήματα καταναλωτών λοιπόν τελικά δεν αντιμετωπίζονται παρκώς και μεγάλη καταναλωτική δύναμη θα μπορούσε να απευθύνεται σε επιχειρήσεις με καλύτερες επιδόσεις. Και όλα αυτά τα χρήματα παραμένουν σε επιχειρήσεις που δεν έχουν καταφέρει να αντιμετωπίσουν σωστά τις διαμαρτυρίες πελατών. Το δεύτερο σημείο στον πίνακα αποτελεσμάτων για τις συνθήκες των καταναλωτών αφορά την ενοποίηση της ελληνικής αγοράς στην Ευρώπη. Γνωρίζουμε ότι αυτό απασχολεί εδώ και πολλά χρόνια την Επιτροπή σα. Τα νέα είναι, θα έλεγα, ανά, ανάμεικτα. Η ηλιανική εσωτερική αγορά απέχει ακόμη πολύ από την πλήρη ενοποίηση. Δεν μας εκπλήσει ίσως το ότι οι καταναλωτές εξακολουθούν να προτιμούν να αγοράζουν προϊόντα και υπηρεσίες στις χώρες τους παρότι παρατηρείται αργή αλλά σταθερή αύξηση στις διασυνοριακές αγορές το 2011. Λοιπόν, σχεδόν ένας στους τρεις Ευρωπαίους αγόρασε προϊόντα ή υπηρεσίες από άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Κατά τα τελευταία πέντε χρόνια σημειώνεται δηλαδή αύξηση της τάξης του 5%. Κινείται δηλαδή πάρα πολύ αργά. Η άλλη πλευρά του νομίσματος είναι ότι οι περισσότεροι λιανοπολιτές ε, προτιμούν να πουλούν προϊόντα και υπηρεσίες σε τοπικούς πελάτες. Οι επιχειρήσεις λοιπόν που δραστηριοποιούνται διασυνοριακά δεν έχουν αλλάξει ιδιαίτερα σε αριθμό από το 2006. Μόνο ένας στους τέσσερις Ευρωπαίους λιανοπολιτές επιλέγει διασυνοριακές ή εξαποστάσεως πωλήσει προς καταναλωτές ε, που διαμένουν σε άλλη χώρα. Εδώ παρατηρούμε επίση ε, σημαντική διαφορά μεταξύ κρατών μελών όπω θα αναμενόταν. Ε, πιο κεντρικέ γεωγραφικά χώρε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι οι χώρε όπου απαντάται περισσότερο, ε, απαντώνται περισσότερε διασυνοριακέ πωλήσει και αγορέ όπω το Λουξεμβούργο για παράδειγμα. Ποια είναι τα εμπόδια που ανησυχούν τους καταναλωτές όσον αφορά την όλη εμπειρία, το κατά πόσο θα φτάσουν τα αγαθά, κατά πόσο θα είναι λατωματικά, τι θα συμβεί σε περίπτωση που πάει κάτι λάθος, η ασφάλεια των συστημάτων πληρωμών και οι λιανοπολιτές ανησυχούν. Βρίσκομαι στη διαφάνεια 13. Εδώ σταματάμε, διαφάνεια 13. Οι λιανοπολιτέ ανησυχούν για τη γλώσσα και για του νόμου προστασίας των καταναλωτών σε άλλα κράτη-μέλη. Επόμενη διαφάνεια, παρακαλώ. Το ηλεκτρονικό εμπόριο θεωρείται πάντοτε πανάκια για την ενοποίηση της λιανικής αγοράς. Έδινε τη δυνατότητα σε μικρές επιχειρήσεις να δραστηριοποιούνται στην εσωτερική αγορά και μείωσε φυσικά τα κόστη και τους φραγμούς συναλλαγών για τους καταναλωτές που ήθελαν να πραγματοποιήσουν αγορές σε άλλα κράτη-μέλη. Το ηλεκτρονικό εμπόριο λοιπόν αυτή τη στιγμή αποτελεί σημαντικό διάβλο για τη λιανική πώληση. Για το λιανικό εμπόριο. Συνολικά τέσσερις από στους 10 Ευρωπαίους καταναλωτές αγόρασαν ε, υπηρεσίες ή προϊόντα online το 2011. Παρατηρείται λοιπόν ε, σταθερή και σχετικά γρήγορη αύξηση συνολικά. Φυσικά θα παρατηρήσετε σημαντικές διαφορές. Ε, το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει αναπτυχθεί περισσότερο στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Σουηδία, τη Δανία, τις κατοχώρες και το Λουξεμβούργο. Και μιλάμε για 70% όλων των καταναλωτών που πραγματοποιούν αγορές online και αυτό πέφτει στο 6% στη Ρουμανία. Όπως αναμένεται υπάρχει ισχυρό συσχετισμός μεταξύ του επίπεδου αγορών online και άλλων δικτών όπως ας πούμε η διάδοση των ευρυζωνικών συνδέσεων. Αυτό επηρεάζει σημαντικά το κατά πόσο επιθ... ενθαρρύνονται οι καταναλωτές να πραγματοποιήσουν αγορές online. Τώρα το χάσμα του ηλεκτρονικού εμπόριου. Το ηλεκτρονικό εμπόριο αυξάνεται σημαντικά. Ε, στόχος είναι του ψηφιακού θεματολογίου το 50% των καταναλωτών να πραγματοποιούν ηλεκτρονικές αγορές μέχρι το 2015. Ωστόσο υπάρχει τεράστια διαφορά μεταξύ του ηλεκτρονικού εμπορίου και του διασυνοριακού εμπορίου. Εάν δείτε λοιπόν ε, η πάνω γραμμή είναι η συνολική ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου σε μπλε χρώμα οι εγχώροι πολιτές είναι η με κόκκινο και οι διασυνοριακοί πολιτές είναι με την κίτρινη γραμμή. Δηλαδή αγορά από πολιτή σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η πράσινη είναι αγορά από πολιτή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει ένα τεράστιο κενό μεταξύ των δύο πάνω και των δύο κάτω ε, γραμμών. Πιστεύουμε ότι αυτό το ο στόχος του 20% ε, είναι, είναι απίθανο να έχει επιτευχθεί μέχρι το 2015. Κρίμα είναι όλα αυτά, γιατί έχουμε πολλά να κερδίσουμε σε ό,τι αφορά χαμηλότερες τιμές και ευρύτερο πλαίσιο επιλογής. Μία από τις μελέτες μας θεωρεί ότι αν φτάσει το στόχο του 15% το ηλεκτρονικό εμπόριο και αν μπορέσουμε να εξαλείψουμε όλα τα προσκόμματα στην ενιαία αγορά, οι καταναλωτές θα κερδίσουν σε επίπεδο ευμάρειας κατά 200 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 1,7 του ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Παρασάγκας απέχουμε όμως προς το παρόν από κάτι τέτοιο. Σημαντικό είναι να θέσουμε και ερωτήματα για το πώς χρησιμοποιούν οι πολίτες το διαδίκτυο αυτή τη στιγμή όχι απλώς για να αγοράσουν, αλλά για να κάνουν έρευνα αγοράς. Αυτό που είναι σαφές είναι ότι ακόμα και αυτοί οι οποίοι εξακολουθούν να αγοράσουν πράγματα από, υλικά, πραγματικά καταστήματα, ψάχνουν στο άειλο ίντερνετ για πολύ καιρό, ψάχνοντας σελίδες, βλέποντας ε, αναφορές οργανώσεων καταναλωτών κτλ. Το επόμενο, η επόμενη διαφάνεια παρακαλώ. Και πάλι, αν κοιτάξετε την ε, κατάσταση που επικρατεί σε διάφορα κράτη-μέλη, βλέπετε να υπάρχει η ίδια τάση. Είναι πιο μεγάλη η διαμεθοριακή ε, αγορά για τις χώρες που είναι πιο μικρές, γιατί όσο πιο μικρή είναι μια χώρα, τόσο πιο μακριά κοιτάζει για να μπορέσει να αγοράσει προϊόντα επιγραμμικά. Οι χώρες οι οποίες έχουν μια μεγάλη και όριμη αγορά στο διαδίκτυο είναι ικανοποιημένε με τις προσφορές που έχουν σε εθνικό επίπεδο. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει υψηλό επίπεδο ηλεκτρονικών αγορών, αλλά ελάχιστοι στο Ηνωμένο Βασίλειο διαλέγουν κάτι από ένα διαδικτυακό τόπο στην Ολλανδία γιατί είναι ικανοποιημένοι μάλλον από αυτά που έχουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αν το συγκρίνουμε όμως με τη Μάλτα και το Λουξεμβούργο, εκεί οι πολίτες θεωρούν ότι <clears throat> είναι καλύτερο να αγοράσουν από ιστότοπους σε άλλα κράτη-μέλη για να έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα επιλογής και καλύτερες τιμές. Στο Λουξεμβούργο είναι κάπως ε, αντίθετα τα πράγματα. Είναι αυτή η ακίδα που βλέπετε στο μέσο της, ε, της διαφάνειας. Υπάρχουν πιο πολλοί που αγοράζουν από το εξωτερικό από ό,τι από το εσωτερικό το επόμενο, η επόμενη διαφάνεια. Ρωτήσαμε λοιπόν τους καταναλωτές γιατί τους αποτρέπει το ηλεκτρονικό εμπόριο και οι διαμεθοριακές αγορές και μας είπαν ότι φοβούνται ότι θα έχουν προβλήματα. Τους ρωτήσαμε επίσης αν είχαν προβλήματα με τις αγορές αυτές. Όπως δείχνουν τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει, υπάρχει πολύ μικρή διαφορά. Αλλά είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα όταν κάνει κανείς διαμεθοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο από ότι εγχώριο εμπόριο, αγοράσει ηλεκτρονικό εμπόριο μέσα στη χώρα του. Είναι καλύτερα να αγοράσει λοιπόν κανείς απ' έξω παρά να αγοράζει από τη χώρα του. Αυτό δεν φαίνεται προφανές. Ένας από τους λόγους είναι ότι αν αγοράσετε από ένα ιστότοπο άλλης χώρας, θα αγοράσετε από μια πιο μεγάλη εταιρεία κατά πάσα πιθανότητα, μια εταιρεία που έχει πιο μεγάλη φήμη και κύρος και αυτό δείχνει γιατί υπάρχει κάποιο μικρό πλεονέκτημα. Ερχόμαστε στο στη λουκούμια διαφάνεια, σχεδόν στην υπολουκούμια. Τι χρειάζεται τώρα να γίνει για να έχουμε καλύτερη ολοκλήρωση της αγοράς λιανικών προϊόντων στον ηλεκτρονικό χώρο. Υπάρχει ένας κατάλογος δράσεων, η οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών που εφαρμόζεται στα κράτη-μέλη. Ξέρω ότι εξετάσετε τις προτάσεις για εναλλακτική επίλυση διαφορών και επιγραμμική ακόμα επίλυση διαφορών. Την πρόταση για ένα ευρωπαϊκό νομοθέτημα σε σχέση με τις αγορές και τις πωλήσει και η πράξη νέας αγοράς υπαριθμών 2, όπου θα αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα προβλήματα. Σας ευχαριστώ, συγγνώμη που μακρηγόρησα, συγγνώμη για τα τεχνικά προβλήματα, αλλά μαζί με τους συναδέλφους μου, που είναι υπεύθυνοι για το συντονισμό του βαθμολογίου, είναι έτοιμοι να απαντήσουν μαζί μου τα ερωτήματά σας. Uh, thank you very much Ευχαριστώ πάρα πολύ, Τζακί. Νομίζω ότι παρακολουθήσαμε πολύ καλά την παρουσίασή σου, γιατί ήταν πολύ καλά διαρθρωμένη και σαφής. Έχουμε τώρα και τις διαφάνειες στα χέρια μας και αντίγραφα του βαθμολογίου. Και εγώ τα έχω παρακολουθήσει με το iPad μου, όπως ίσως και άλλοι τύποι. Αγαπητοί συνάδελφοι, φαντάζομαι ότι έχετε κάποια ερωτήματα η κυρία Πιετικάινεν είναι η πρώτη αντιπρόεδρός μας και θέλει να λάβει το λόγο για τα θέματα αυτά. Επίσης ο κύριος Σφάμπ εξεδήλωσε τη θέλησή του να λάβει το λόγο. Ξεκινάμε με αυτούς τους δύο μιλητές. Σύρπα. Ευχαριστώ. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πλήρη, την ε, ε, εξονυχιστική σας παρουσίαση των διαφορών σημείων. Νομίζω ότι μας δίνει μια πολύ καλή εικόνα και τροφή για σκέψη. Θέλω να σας ευχαριστήσω λοιπόν για τις ε, έρευνες αυτές που κάνετε μαζί με τα κέντρα καταναλωτών. Θα ήθελα να γύρω τρία ζητήματα σε σχέση με τις μελλοντικές εξελίξεις στον τομέα αυτό. Κάτι το οποίο δεν χρειάζεται να το ασχολήσω είναι ότι και εγώ ήδη έχω κάποιες αμφιβολίες ότι η κοινή νομοθεσία για τις αγορές σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα επιτύχει κάποιο θετικό αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά την εναρμόνιση της αγοράς και σε ό,τι αφορά την σαφήνεια για τα προαπαιτούμενα για την προστασία των καταναλωτών. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να έχουμε όλοι υπόψη μας. Επίσης όμως θα ήθελα να ακούσω και τα σχόλια για τις μελλοντικέ πρωτοβουλίες και για το ρόλο των κέντρων καταναλωτή. Και πρόκειται για τρία θέματα. Ξέρουμε ότι λειτουργούν διαφορετικά τα... σε διάφορα κάτι μέλη και επομένω αυτό επηρεάζει το τελικό αποτέλεσμα. Θα ήθελα να ακούσω και κάποιες απόψεις για το πώς τα κέντρα αυτά θα μπορούσαν να ενισχυθούν με ευρωπαϊκή προοπτική δηλαδή να έχουν περισσότερους πόρους, να αντιμετωπίσουν καλύτερα τη γραφειοκρατία. Ένα άλλο θέμα να είναι η εναλλακτική επίλυση διαφορών, ADR. Εγώ, επειδή έρχομαι από τη Φιλανδία, ξέρω ότι έχουμε ένα καλό ιστορικό για τα θέματα αυτά και μου φαίνεται πολύ θετική η ιδέα ότι τα κέντρα καταναλωτών μπορούν να διαδραματίσουν ένα πιο ισχυρό και επίσημο ρόλο για την ε, εναλλακτική ε, επίλυση διαφορών στο μέλλον και θα ήθελα να έχω και τα σχόλια σας για το θέμα αυτό. Τέλος, αλλά δεν είναι το, το λιγότερο σημαντικό γιατί ξέρετε ότι είμαι συντάκτρια της γνωμοδότησης για τα δικαιώματα των επιβατών. Έχουμε εκθέσεις από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κέντρο Καταναλωτών ότι πάνω από το 1, από το 33,3 των παραπώνων αφορούν θέματα εισιτηρίων αεροπορικών εταιριών και θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο να ξέρουμε πώς μπορεί να υπάρξει μεγαλύτερη ενίσχυση αυτών των κέντρων εκεί και να παίξουν τα κέντρα καταναλωτών περισσότερο το ρόλο του εστιακού σημείου σε σχέση με τις κρατήσεις εισιτηρίων κτλ. Αν μπορούν να το αναλάβουν αυτό. Ευχαριστώ, σας είπα, ο Ανδρέας Σφάμπ. Ευχαριστώ. Λοιπόν που καθυστέρησα, ήμουν στην Οικονομική Επιτροπή και συζητούσαμε άλλη οδηγία για την οποία είναι συναρμόδια για γνωμοδότηση η Επιτροπή μας. Ποια είναι τα θετικά του βαρομέτρου. Υπάρχουν μερικές επιφυλάξεις συνολικά για το θέμα του βαρομέτρου, ωστόσο υπάρχουν τέσσερα θέματα που μας δείχνουν καθαρά τι μπορούμε να κάνουμε με τα αποτελέσματα αυτών των ε, δημοσκοπήσεων. Πρώτο, το βαρόμετρο επιβεβαιώνει ότι το εμπόριο μέσω διαδικτύου ενισχύεται, κυρίως όμως στο εσωτερικό των χωρών, παρόλο που υπάρχει σημαντική δυνατότητα εξοικονομήσεων για τους καταναλωτές εάν κάνουν και διεθνείς συναλλαγές. Τώρα, διαφάνεια 17, το δείχνει καθαρά. Πρέπει να ρωτήσουμε περισσότερο τι μπορεί να βελτιωθεί σε ό,τι αφορά την παράδοση των εμπορευμάτων, διότι πολλοί καταναλωτές εκφράζουν φόβους ότι η παράδοση ή δεν γίνεται καθόλου, είτε το εμπόρευμα υφίσταται βλάβες, είτε καθυστερεί. Τώρα, η κυρία Κέπχατ βλέπω κυρια κεμχατ βλεπω εφυγε αλλά αυτή η delivery είναι πολύ κρίσιμος παράγοντας, αυτή η παράδοση του εμπορευματο. Χαίρομαι που υπάρχει τώρα η πράσινη βίβλο για, το, για την ε, παράδοση εμπορευμάτων, ή δεμάτων. Αλλά αυτό δεν μπορεί να επιλύσει το πρόβλημα αυτό και αυτό είναι κάτι το οποίο εναπόκειται στα εθνικά συστήματα. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε αν δεν επιλύσουμε το θέμα αυτό. Ένα δεύτερο σημείο όπως είπε και ο κύριος Σαρίας στην ε, πρόταση πρωτοβουλίας του, ένα σημαντικό θέμα. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι ότι οι γνώσει των καταναλωτών για τα δικαιώματά τους είναι πολύ περιορισμένη. Και γι' αυτό η οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών θα παίξει ένα σημαντικό ρόλο να καθορίσει κοινού κανόνες σε όλα τα κράτη-μέλη για να υπάρξει εδραίωση των δικαιωμάτων των καταναλωτών θεωρούμε ότι μπορούμε να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο αυτή την ενημέρωση των καταναλωτών. Γνωρίζω ότι η οδηγία ακριβώς και στους τομείς όπου θα φέρει πλήρη εναρμόνιση, ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις δεν θα εφαρμοστεί με ομοιόμορφο τρόπο. Τι κάνει λοιπόν η Κομισιόν. Η Κομισιόν τελικά προ προωθεί την πλήρη εναρμόνιση για λόγους επαγγελματικής ανέλυξης και μόνο και δεν ενδιαφέρεται για την ε, εφαρμογή αυτών των οδηγίων, έκανα και μια προφορική ερώτηση προς την κυρία Ρέντινγκ. Θεωρώ ότι αυτό δεν είναι σωστό. Και πρέπει να σκεφτούμε και την οδηγία για τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές. Όπως λέει το Ευρωβαρόμετρο, ότι εξακολουθούμε μετά από 7 χρόνια να αντιμετωπίσουμε πολιτικές οι οποίες είναι αθέμητες, ακόμα και σε περιπτώσεις που υπάρχει πλήρης εναρμόνιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχει απαγόρευση τέτοιου είδους πρακτικών. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν δίνει την πρέπουσα προσοχή στην εφαρμογή παλιότερων οδηγιών και μόνο νοιάζεται να φέρνει νέες προτάσεις. Κύριε Μάνερ, λοιπόν, στον τομέα αυτό που βλέπετε να υπάρχει πλήρης εναρμόνιση, να υπάρχει καλύτερη εφαρμογή ή παραμένουμε σε ένα επίπεδο άνησης εφαρμογής σε ό,τι αφορά τον καταναλωτή. Δεν θέλω λοιπόν να περάσω σε περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά από ό,τι γνωρίζουμε λοιπόν είναι φανερό ότι δεν γνωρίζουν τα δικαιώματα τους ακόμα οι καταναλωτές και επομένως δεν μπορώ να δω τι θα προκύψει από μια πλήρη εναρμόνιση. Τέλος. Έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα αυτό το ευρωβαρόμετρο σε σχέση με τα θέματα αυτά για την εφαρμογή αυτών των οδηγιών σε σχέση με άλλα θέματα με τους καταναλωτές. Το γεγονός ότι έχει ξεκινήσει με συστάσεις οι οποίες είναι ειδικέ για κάθε χώρα, χωρίς να φτάνει στο επίπεδο πάντα του να επωνυδίζει τις χώρες αυτές, ώστε να υπάρχει μια μεγαλύτερη σαφήνεια σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται τα δικαιώματα των καταναλωτών σε κάθε χώρα και δεν έχουμε μονάχα μια γενική εντύπωση για το τι γίνεται στην ενιαία αγορά. Αυτό το βρίσκω ότι είναι πάρα πολύ θετικό Δεν συμφωνώ πάντα με αυτά τα οποία, δεν είναι πάντα ευχάριστα αυτά τα οποία παίρνουμε από το ευρωμαρώματο, αλλά είναι σημαντικό το ότι έχουμε καταχώρες ε, συστάσεις και συμπεράσματα και αυτό μας βοηθάει να προχωρήσουμε πολύ περισσότερο στην εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων. Ευχαριστώ. Η κυρία Ρόιτοβα. Σας ευχαριστώ. Δεν θέλω να επαναλάβω αυτά που ελέγχθησαν ήδη. Θέλω να προσθέσω λίγα, απλώς υπογραμμίζοντας αυτά τα οποία ελέγχθησαν προηγουμένως. Η εμπιστοσύνη στην ασφάλεια των αγαθών και στις σωστές νομικές διασφαλίσεις, αυτά είναι δύο πράγματα τα οποία είναι αλληλένδετα. Και επίσης συνδυάζονται με την εμπιστοσύνη για την ε, λειτουργία της δημοκρατίας και όχι μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει ένας κίνδυνος ο οποίος ε, υπάρχει σε ορισμένα κράτη-μέλη, μεταξύ των οποίων και στη δική μου χώρα, που είναι το ότι υποτιμούμε το ρόλο της προστασίας των καταναλωτών. Σε πολλές χώρες είναι το Υπουργείο Εσωτερικών που ασχολείται με τα θέματα. Αλλά σε άλλες περιπτώσεις είναι οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εμπορίου που ασχολούνται με τα θέματα αυτά, αλλά παρατηρούμε πολλές φορές ότι δεν υπάρχει συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων αρχών. Στη χώρα μου υπάρχουν διάφορες εποπτικές αρχές που λένε πάντα ότι δεν είναι η αρμοδιότητά τους να ασχοληθούν με το θέμα αυτό και πετάνε τον παλάκι σε κάποιον άλλο φορέα. Σε κτηνιατρικές αρχές, σε αρχές τηλεπικοινωνίας. Ως εκ τούτου, το σύστημα είναι τόσο κατακαιρματισμένο ώστε εκτός αν υπάρξει μια κατακραυγή από τα μέσα ενημέρωσης ή κάποια εκστρατεία αυτού του είδους, όλα αυτά τα θέματα απλώς θα παραγνωρίζουν οι αρμόδιοι φορείς. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω την Κομισιόν κατά πόσο θα μπορούσε να ελέγξει με ποιο τρόπο και σε ποιο βαθμό τα κράτη-μέλη παίρνουν στα σοβαρά τις καταστάσεις αυτές και αναφέρομαι κυρίως στα κράτη-μέλη τα οποία δεν είχαν τόσο καλή βαθμολογία στο βαθμολόγιο, τι κάνουν για να αντιμετωπίσουν το θέμα της προστασίας των καταναλωτών και ιδίως σε ποιο βαθμό επιζητούν να εξασφαλίσουν καλύτερο συντονισμό και καλύτερη συνεργασία των ανεξαρτήτων εποπτικών αρχών για τα θέματα αυτά και να εναρμονίσουν την αντιμετώπιση του. Ευχαριστώ. Κανείς άλλος? Άλλος, άλλος κανείς επιθυμεί να σχολιάσει. Καλά, λίγα δικά μου τότε. Πολλά δεδομένα εδώ και τονίσατε ορισμένα. Πολλά δεδομένα επίσης σχετικά με την επιβολή για τους προϋπολογισμούς. Ίσως την επόμενη φορά μετά από την έκκληση του Ανδρέα Σφάπ θα είναι ενδιαφέρον να τα έχουμε τα δεδομένα αυτά γιατί είναι σημαντικά για το έργο μας κυρίως για τις ε, εμπορικές πρακτικές που ξέρουμε ότι πρόκειται να υποβάλλεται θεωρημένη πρόταση σύντομα. Έρχομαι τώρα σε κάτι που είπε η κυρία Πιετικάινεν για εργαλεία που μας απασχολούν τώρα. Για παράδειγμα, οι ανησυχίες των καταναλωτών για τις αγορές στο διαδίκτυο που τους απασχολούν κυρίως θέματα παράδοσης είτε καθυστέρηση είτε ζημιέ ζημιές που όλα αυτά είναι σημαντικά και υποσκάπτουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Δεν είναι μόνο ότι οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους. Και η έκθεση της digital Markets είναι σημαντική γιατί έβαλε όλα αυτά τα πράγματα σε ένα ενίο σύνολο. Εγώ νομίζω πάντως, διότι είχαμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση για την ε, μελέτη αντικτύπου του Common Sales Law και νομίζω ότι έχει εδώ πλήθος δεδομένων πολύ μεγαλύτερο που θα πρέπει να περάσουν τελικά στο σύστημα. Ζητήσαμε από την μονάδα που κάνει τις μελέτες αντικτύπου να τα εξετάσει και να συνεργαστούμε μαζί σας για να δούμε ορισμένα από τα θέματα αυτά. Και το δεύτερο θέμα έχει σχέση με αυτά. Δηλαδή, μιλώ για τον δίκτυ και τις γνώσεις των καταναλωτών και των λιανοπολιτών. Και διαρωτώ με αν μπορείτε να μας εξηγήσετε. Φαίνεται να υπάρχει περιορισμένο σχημα... Ε, συσχετισμός ανάμεσα στην εμπιστοσύνη και στη γνώση των δικαιωμάτων. Λουξεμβούργο και Ενωμένο Βασίλειο είναι ε, ε επικεφαλής του καταλόγου σας ό,τι αφορά την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Αλλά για, την εμπιστοσύνη, ενώ για τις γνώσεις είναι στο τέλος του καταλόγου, κάτω-κάτω. Πώς λοιπόν αντιμετωπίζουμε τα θέματα των καταναλωτών στο επίπεδο της πολιτικής, αυτό δείχνει και βέβαια μας απασχολούν θέματα εμπιστοσύνης καταναλωτών, αλλά αυτό που ενδιαφέρει τους καταναλωτές είναι να, πάρουν, να παραλάβουν το αντικείμενο που ε, παρήγγειλαν έγκαιρα και ασφαλώς. Είναι σημαντικό να εξεταστεί αυτός ο συσχετισμός δηλαδή και σε σχέση με την αντίληψη που έχει ο κόσμος για την ασφάλεια των προϊόντων και την εμπιστοσύνη ότι υπάρχει ένα σύστημα δηλαδή το οποίο ασχολείται με την ασφάλεια των προϊόντων. Μιλούμε για τα δικαιώματα των καταναλωτών. Άλλη μια οδηγία έχουμε εδώ τώρα, το δίκαιο δηλαδή των πωλήσεων και για να βελτιωθεί το σύστημα θα πρέπει να βελτιωθεί σε ένα ενίο σύστημα αντί να έχουμε 28 διαφορετικά και αυτό θα οδηγήσει σε βελτίωση εμπιστοσύνη καταναλωτών. Απάντηση Κομισιόν. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στα σχόλιά σας όσο μπορώ. Πρώτα απ' όλα, κυρία Πιετακάινεν, και τα σχόλια της όσον αφορά τα ευρωπαϊκά κέντρα καταναλωτών. Φαντάζομαι ότι αναφέρεστε απευθείας στα ευρωπαϊκά κέντρα καταναλωτών και όχι στους οργανισμούς γενικότερα. Έχουμε, όπως γνωρίζετε, στο πρόγραμμα για τους καταναλωτές, που είναι ουσιαστικά το πρόγραμμα χρηματοδότησης για το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο από το 2014. Το πολιετές έχουμε αλλάξει τους κανόνες υποστήριξης των ECC των Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτών ώστε να λαμβάνουν περισσότερη χρηματοδότηση. Προς το παρόν είναι 50-50 μεταξύ εμάς και των κρατών μελών και θα το αλλάξουμε τώρα σε 70% συμμετοχή της Κομισιόν. Ελπίζουμε ότι δεν θα μειώσουν τα κράτη-μέλη τα κράτη-μέλη το ποσά που καταβάλουν ε, έτσι ώστε να αυξηθεί η χρηματοδότηση των Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτών και η αλήθεια είναι ότι τα καλύτερα τέτοια κέντρα ECC επιτελούν μια πολύ ωφέλιμη λειτουργία, δημιουργούν εμπιστοσύνη στις διασυνοριακές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά. Τα καλύτερα ECC και το Βέλγιο αποτελεί ένα άριστο ε, παράδειγμα ε, παρέχει δυνατότητες στους καταναλωτές μέσω ενημέρωσης ε, για την εσωτερική αγορά και θα ήθελα και άλλα ίσως να ακολουθήσουν αυτό το παράδειγμα. Προσπαθούμε αυτή τη στιγμή μέσω των εργασιών μας να διαδώσουμε τις καλύτερες πρακτικές μέσα στο δίκτυο όσον αφορά τις ίσεις για τα ODR και τα EDR. Είμαστε βεβαίω ανοιχτοί για αυτό και φυσικά πολλά συζητώνται όσον αφορά την εκτίμηση της κυρίας Τούν για τις πλατφόρμες ODR, όσον αφορά τον ρόλο που θα μπορούσαν να επιτελέσουν τα ECC. Εμείς είμαστε διατεθειμένοι να εξετάσουμε το ενδεχόμενο ενό ενισχυμένου ρόλου. Γνωρίζουμε ότι σήμερα Υπάρχουν περιπτώσεις όπου τα ECC δεν κατάφεραν να επιλύσουν με δική τους διαμεσολάβηση μέσω του καταναλωτή και του λιανοπολιτή ή μέσω για τις διενέξεις μεταξύ καταναλωτών ε, και λιανοπολιτών στο 10% των περιπτώσεων βρίσκουν εναλλακτική επίλυση διαφορών. Συνεπώς μόνο μία στις δέκα περιπτώσεις ε, καταλήγει σε μία επαρκή λύση ADR ε εναλλακτική επίλυση διαφορών. Θεωρούμε λοιπόν ότι οι προτάσεις που γίνονται θα βελτιώσουν αυτή την κατάσταση, αλλά θα πρέπει να βασιστούμε στην υπάρχουσα εμπειρία των Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτών. Όσον αφορά τα δικαιώματα των επιβατών ε, αεροπορικών εταιριών, έχετε δίκιο. Διαβάζοντα τα στοιχεία κάθε χρόνο, οι μεταφορές είναι ο τομέας όπου υπάρχουν τα περισσότερα παράπονα στο ECC. Και όταν μιλάμε μεταφορέ, μιλάμε κυρίω για αερομεταφορέ. Οι αερομεταφορέ παρουσιάζουν τα περισσότερα προβλήματα. Δεν αφορά μόνο τα δικαιώματα των επιβατών με την έννοια της, του κανονισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε και τι εισαπολιστή τη αποσκευέ ε, που ανήκουν στην ίδια κατηγορία. Συνεργαζόμαστε στενά με του συναδέλφου στην Γενική Διευθυνσή μου, ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι οι τελευταίε και πιο ενημερωμένε πληροφορίε διαδίδονται στο δίκτυο των ECC. Αν υπάρχει νέα νομολογία, για παράδειγμα, ενημερώνουμε τα ECC. Επίσης προσπαθούμε τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Καταναλωτών να έρθουν πιο κοντά στα, ε, στους εθνικούς φορείς επιβολής του νόμου όσον αφορά τον κανονισμό για τους επιβατές ενέργειων μεταφορών. Ενημερωτικά 4 Ιουλίου φέτος, ε, η ημερομηνία που επελέγει κατά τύχη, θα διοργανωθεί μια ημερομηνία ε, επιβατών αεροπορικών εταιριών σε μεγάλα αεροδρόμια της Ευρώπης, όπου τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Καταναλωτών θα συνεργάζονται με αεροδρόμια, τοπικές αρχές επιβολής του νόμου για την κοινοποίηση, την ενημέρωση του κοινού όσον αφορά τα δικαιώματα των επιβατών. Ε, φυσικά αυτό γίνεται ήδη στα αεροδρόμια, αλλά τώρα θα έχουμε πραγματικούς ανθρώπους επιτόπου οι οποίοι θα ενημερώνουν τον κόσμο στις αρχές των καλοκαιρινών διακοπών. Συμφωνώ απόλυτα με όσα ε, είπατε, όσα όταν μιλήσαμε με τους λιανοπολιτές. Όχι γι' αυτό, αλλά στο πλαίσιο μελετών μας Μία από τις αιτίε που μας έδωσαν ε, για να μην επεκτείνουν τις πωλήσει τους διασυνοριακά ήταν ότι θεωρούσαν ότι δεν μπορούσαν να εξασφαλίσουν επαρκές επίπεδο εξυπηρέτησης για τους ε, πελάτες τους. Για παράδειγμα, ταχυδρομικέ υπηρεσίε σε άλλε χώρε που δεν ήταν επαρκού ποιότητα ε, και προτιμούσαν σε αυτή την περίπτωση οι πολιτέ να μην μπουν στην αγορά αντί να μπουν παρέχοντας ε, ανεπαρκή εξυπηρέτηση. Θεωρούμε λοιπόν ότι η παράδοση των δεμάτων θα πρέπει να γίνεται σωστά και οι συναδελφοί μας στην ε, Γενική Διεύθυνση ΜΑΚΤ ε, εργάζονται προς αυτή την κατεύθυνση. Η τώρα ευαισθητοποίηση, τα δικαιώματα μάλλον και θα επανέλθω στο σημείο του Προέδρου στο τέλος του χρόνου θα συνεργαστούμε με τους συναδέλφους της Γενικής Διευθύνσης Δικαιοσύνη για κάποιες περισσότερες εκστρατείες. Πιστεύω ότι οι πληροφορίες του πίνακα αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές είναι σημαντικές, διότι εδώ μιλάμε για ε, δράσεις μεταβλητής γεωμετρίας. Δεν έχει νόημα να βελτιώσουμε τη γνώση των καταναλωτών στις χώρες όπου ήδη είναι υψηλή. Θα πρέπει να επικεντρώσουμε τις προσπαθίες μας στις χώρες όπου παρατηρούνται οι λήψεις. Αυτό που επίσης κάναμε, και αυτό αφορά το σημείο της πλήρους αναρμόνισης, είναι προσπαθούμε να συνεργαστούμε με ένα δίκτυο συνεργασίας για την προστασία των καταναλωτών, δίκτυο το οποίο συγκεντρώνει όλες τις αρχές επιβολής του νόμου, τις δημόσιες αρχές επιβολής του νόμου, ώστε να ερμηνεύεται όσο το δυνατόν με πιο κοινό τρόπο η νομοθεσία τόσο όσον αφορά τις αθέμητες πρακτικές, όσον αφορά τους όρους των συμβουλέων και σύντομα και η οδηγία δικαιωμάτων των καταναλωτών διοργανώνουν τώρα πολλά εργαστήρια που μελετούν συγκεκριμένε ε, υποθέσει, ε, προσπαθούν να συμφωνήσουν για τον τρόπο χειρισμού του. Έχουμε εργαστήρια όπου συγκεκριμένοι τομεί ε, θέμη του ανταγωνισμού συζητώνται ώστε να υπάρξει ανταλλαγή πληροφοριών σε θέματα εντοπισμού, έρευνας, δίωξης αθέμητων εμπόρων στην αγορά είναι ένα σημείο στο οποίο, θα, όπως αναφέρετε πολύ σωστά, θα πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε. Κύριε Ρόιτερ, αναφέρατε την εμπιστοσύνη στη λειτουργία της αγοράς και ότι αυτή αποτελεί ένα απόσπαστο κομμάτι της εμπιστοσύνης στη συνολική λειτουργία μιας δημοκρατικής χώρας και μιας χώρας γενικότερα. Και πάλι συμφωνούμε μαζί σας. Ο κατακαιρματισμός μεταξύ διαφόρων φορέων πιστεύω ότι είναι ένα από τα προβλήματα. Ορισμένες χώρες το έχουν ξεπεράσει. Κοιτώντας τις κατοχώρες ετοιμάζονται να διοργανώσουν μια υπερρυθμιστική αρχή για τις τηλεπικοινωνίες, τους καταναλωτές, την ενέργεια και νομίζω τα ύδατα. Δηλαδή συγκεντρώνουν όλες αυτές τις λειτουργίες σε έναν ενιαίο οργανισμό. Αυτό που κάνουμε λοιπόν εμείς ε, και πάλι στο πλαίσιο του δικτύου πολιτικής καταναλωτών, δηλαδή τα Υπουργεία Προστασίας των Καταναλωτών, προσπαθούμε να μοιραστούμε αυτή την εμπειρία. Λειτουργεί αυτή η συγκέντρωση όλων των ρυθμιστικών αρχών ή μήπως υπάρχουν άλλοι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να διασφαλίσουμε το συντονισμό τους. Επίσης, ε, συνεργαζόμαστε με το ΜΠΕΟΚ, e τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Καταναλωτών, Όσον αφορά το κίνημα των καταναλωτών στις νοτιοανατολικές χώρες, οι χώρες AC όπως αναφέρονται, ένα κίνημα καταναλωτών δεν λαμβάνει μορφή μέσα σε μια μέρα φυσικά. Εδώ μιλάμε στις βόρειο-δυτικές χώρες. Φυσικά το κίνημα καταναλωτών ξεκίνησε πριν από 50, 60, 70 χρόνια, ενώ σε άλλες χώρες αποτελεί ακόμη σχετικά νέο κίνημα. Πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσουμε να πείθουμε τις δημόσιες αρχές και όσους χαράσουν πολιτική ότι η ισχυρή φωνή των καταναλωτών δεν είναι επιβλαβής για τις επιχειρήσεις. Αντιθέτως, η ενδυνάμωση και η παροχή γνώσεων στους καταναλωτές βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα, κάνει πιο ικανές τις επιχειρήσεις, βελτιώνει τον ανταγωνισμό, διασφαλίζει ότι ανταποκρίνονται σωστά οι επιχειρήσεις στις απαιτήσεις της αγοράς τέλος το σημείο που ανέφερε ο, ο πρόεδρος η επιβολή θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με προσοχή κάποια κράτη-μέλη δυσκολεύτηκαν στη συγκέντρωση των στοιχείων. Δεν υπάρχει καμία διασφάλιση ότι τα στοιχεία και ο δείκτης αυτός είναι πλήρης και εξατλητικός, αλλά είναι ό,τι καλύτερο έχουμε αυτή τη στιγμή. Ο συσχετισμός μεταξύ της γνώσης των δικαιωμάτων των καταναλωτών από τους ίδιους καταναλωτές και την εμπιστοσύνη Πιστεύω μπορούμε να δημιουργήσουμε και άλλους συσχετισμούς για σας. Δεν είναι πρόβλημα αυτό, είναι αρκετά εύκολο. Είναι ενδιαφέρον πιστεύω ότι οι αγορές εκείνες που, τις οποίες οι καταναλωτές θεωρούν πιο άνετες, όπου νιώθουν πιο ασφαλείς οι καταναλωτές και σωστά προστατευμένοι, δεν είναι απαραίτητα οι αγορές όπου, για τις οποίες οι καταναλωτές γνωρίζουν λεπτομερώς τα δικαιώματά τους. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που θα έπρεπε ίσως να εξετάσουμε. Ίσως η εμπιστοσύνη θα πρέπει να, να, έχει περισσότερο βάρος από τη γνώση. Όταν γνωρίζεις ότι ένας λιανοπολιτής θα σεβαστεί τα δικαιώματά σου, ε, δεν χρειάζεται να γνωρίζεις τις λεπτομέρειες. εφόσον υπάρχει επαρκή πίεση εντό τη αγορά να συμπεριφερθούν σωστά, τότε οι καταναλωτέ ανασυχούν λιγότερο. Δεν ασχολούνται ιδιαίτερα με το να γνωρίζουν λεπτομερώ τα δικαιώματά του και αυτό θα μπορούσαμε να το ερευνήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ και πάλι που μα δώσατε όλα αυτά τα στοιχεία, λέει ο πρόεδρο. Υπάρχει μια άλλη πτυχή την οποία δεν θίξαμε. Επειδή ασχολούμεθα αυτή τη στιγμή και με το πρόγραμμα των καταναλωτών είναι το θέμα της ε, δημιουργίας οργανώσεων καταναλωτών. Και βλέπω εδώ ότι από την έκθεσή σας υπάρχει μεγάλος συσχετισμός με την, μεταξύ της κατάστασης των καταναλωτών και της εμπιστοσύνης τους οι ε, φορείς καταναλωτών που υπάρχουν. Ναι, θα μπορούσατε να δείτε περισσότερες ε, ε, περισσότερους συσχετισμούς. Δεν καλύψατε ίσως για λόγους αυροφροσύνης αυτά τα οποία σας ε, ζήτησα, αλλά ίσως αν δείτε το θέμα της εμπιστοσύνης στους φορείς καταναλωτών <clears throat> θα βρείτε κάποια καινούργια στοιχεία και εμείς πιέσαμε τους εκπροσώπους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 είναι το θέμα του ποιος στο μέλλον θα πρέπει να αντιμετωπίζει γενικά τα θέματα προστασίας των δικαιωμάτων των επιβατών. <clears throat> Και για μένα, παρά το γεγονός ότι αυτά τα δικαιώματα είναι τμήμα των δικαιωμάτων των καταναλωτών, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με ειδικό τρόπο, ιδίως στο μέλλον, όταν έχουμε ένα συμπιλημένο κατάλογο δικαιωμάτων που θα βρίσκεται σε μία οδηγία να τα έχουμε στην αρμοδιότητα της δικής μας Επιτροπής που θα πρέπει να επιληφθεί των μελλοντικών ενεργειών για τα θέματα αυτά. Και έχουμε συζητήσει το θέμα αυτό και με τους σκιώδεις εισηγητές σε σχέση με την <clears throat> αρμοδιότητα της Επιτροπής μας σε αυτά τα θέματα. Λοιπόν, οι βασικές σκέψεις τώρα στο θέμα αυτό. Όπως ξέρετε και με άλλα δικαιώματα καταναλωτών υπάρχουν τεράστιες πολυπικιλίε διαφορές και χάσματα μεταξύ των κρατών μελών, μεταξύ διαφορών, διαφορών τρόπων μεταφοράς και ιδίως μεταξύ μεταφορικών ε, μεταφορών που είναι διαμεθοριακού χαρακτήρα. Γι' αυτό είναι σημαντικό να έχουμε ένα μονάχα συγκεκριμένο πλαίσιο που να καλύπτει όλες τις ρυθμίσεις για τα δικαιώματα των επιβατών και να μειώσουμε τον κατακαιρματισμό και την έλλειψη συνοχής του πλαισίου που υπάρχει τώρα. Να έχουμε ένα πλαίσιο το οποίο θα εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη-μέλη, σε όλες τις μορφές μεταφορών και κυρίως τις διαμεθοριακές μεταφορές, όπως πολύ σωστά τόνισε και η Κομισιόν, τα δικαιώματα των επιβατών θα πρέπει να λαμβάνονται πλήρως υπόψη σε όλα τα κρατη και για όλους τους τρόπους μεταφοράς. Έχουμε επίσης τα θέματα για την πρόληψη των διακρίσεων και την παροχή πληροφοριών. Και υπάρχουν και πολλά θέματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε, όπως ελέγχθη προηγουμένως, γιατί είπα ότι ένα τρίτο των παραπώνων για τους ε, για θέματα καταναλωτών έρχονται από προβλήματα μεταφορών. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει πληροφόρηση για όλους τους καταναλωτές προτού αγοράσουν κάποια ταξιδιωτικού χαρακτήρα υπηρεσία και να υπάρχει βοήθεια σε όλα τα στάδια του, της μεταφοράς τους. Τρία θέματα τώρα τα οποία ζητούν περισσότερη προσοχή μας στο μέλλον. Οι πολυτροπικές μεταφορές. Ξέρουμε ότι τα μεγαλύτερα προβλήματα εμφανίζονται όταν εμπλέκονται διαφορετικές μορφές μεταφορών και από, μέσα σε πολλά κράτη-μέλη. Παίρνετε ένα αεροπλάνο, ένα τρένο και ένα λεωφορείο και περνάτε δύο-τρία κράτη-μέλη. Και κάτι πάει στραβά σε αυτή την αλλαγή μέσων μεταφοράς και το ερώτημα είναι ποιος είναι ο αρμόδιος για να ασφαλίσει και να δώσει αποζημίωση για τα θέματα αυτά και τι είδους εγγύηση έχουμε ότι θα λειτουργήσουν με σωστό τρόπο αυτές οι ενέργειες μεταφοράς και θα τύχουν σεβασμού τα δικαιώματα των μεταφερομένων. Και εδώ είναι το θέμα του τι θα μπορούσαν να κάνουν τα ευρωπαϊκά και τα καταναλωτών για το ζήτημα αυτό θα έπρεπε να αναπτύξουμε περαιτέρω στοιχεία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για να βελτιστοποιήσουμε την διατροπική μεταφορά. Γιατί είναι πολύ δύσκολο όλα αυτά να τεθούν σε επίπεδο ευθύνης των μεταφορέων και στην εθελοντική του συνεργασία. Όσο πιο πολύ ταξιδεύουμε, τόσο πιο πολύ εσωτερική αγορά θέλουμε, όσο πιο πολύ εσωτερική αγορά θέλουμε, τόσο μεγαλύτερη ελευθερία διακίνηση των πολιτών μας θέλουμε και επομένως έχουμε ένα πλέγμα προβλημάτων που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Και τουλάχιστον από την έποψη της παροχής πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήταν χρήσιμο να έχουμε μία ενιαία ιστοσελίδα. Ένα δεύτερο που να δίνει πληροφορίες. Δεύτερο θέμα είναι το θέμα των παραπώνων. Φυσικά, σε κάθε τερματικό σταθμό, σε κάθε αεροδρόμιο θα πρέπει να υπάρχει ένα γραφείο παραπώνων αλλά τίθεται το ερώτημα και έθεσα το ερώτημα στην Κομισιόν προηγουμένως. Πώς θα διευκολύνουμε ιδιαίτερα σε αυτές τις περιπτώσεις που είναι πολυτροπική η μεταφορά. Πώς θα μπορούσαμε να διευκολύνουμε την πρόσβαση των επιβατών και την κατάθεση παραπώνων. Σε ποιον θα πρέπει να απευθυνθούν. Τέλος, έχουμε τους επιβάτες με περιορισμένη κινητικότητα. και τα άτομα που έχουν αναπηρίες, τα ηλικιωμένα άτομα που χρειάζονται βοήθεια. Πρέπει να έχουμε μια ολιστική προσέγγιση για όλους αυτούς. Και όταν είναι και πολυτροπική μεταφορά ατόμων που είναι ανάπηροι αλλά και ηλικιωμένοι και χρειάζονται και βοήθεια, τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Α, σε δέαμα πηγαίνουμε από ένα κράτος μέλος στο άλλο. Εκεί γίνεται χαμός. Επομένως χρειαζόμαστε πανευρωπαϊκά εργαλεία για να μπορέσουμε να δίνουμε τις καλύτερες δυνατές πληροφορίες στα άτομα αυτά τα οποία μπορεί να είναι ανάπηρα, ηλικιωμένα και τα δύο για την ανάγκη να έχουν υποστήριξη και βοήθεια από το σπίτι τους μέχρι το άλλο μέρος στο οποίο πηγαίνουν, το τελικό του προορισμό. Και υπάρχουν και άλλα θέματα αν υπάρξει επίσης κάποια αλλαγή σε σχέση με, τις, ε, με τα πακέτα ταξιδίου, με το δικαίωμα καταγγελίας μιας τέτοιας σύμβασης για ταξίδι και το τρόπο υποβολής σε παραπών. Δεν θα τα πω όλα αυτά, αλλά μπορούμε να επανέλθουμε. Σας ευχαριστώ, λέει και ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μάντερς αντιμετωπίζει κάποιο, κάποια πίεση χρόνου. Ε, ναι, κυρία Χέντε, να του δώσω πρώτο το λόγο. Συμφωνεί, συμφωνεί. Της παραχωρεί τη θέση Ναι, έχω μια συζήτηση ε, στο ραδιόφωνο. Θα διαβάσω λοιπόν τα σχόλια που κάνει η κυρία Παρβάνοβα, η οποία ευχαριστεί την κυρία είναι για το σχέδιο γνωμοδοτήσεως. Η κυρία Παρβάνοβα χαίρεται που ορισμένες από τις ιδέες που πρότεινε μπαίνουν στην γνωμοδότηση για τα δικαιώματα των επιβατών, για τα οποία ήταν ε, ε, αρμοδία Ένα, μια πτυχή που θα ήθελε να τονίσει ιδιαίτερα η κυρία Παρβάνοβα ε, είναι η διαφάνεια των τιμών και ιδίω για τους ναύλους με κρυφό κόστος, για παράδειγμα όταν χρησιμοποιείται πιστοτική κάρτα και θα πρέπει η τελική τιμή του ναύλου να, είναι, να ταποκρίνεται στο πραγματικό κόστος. Και επίσης να προστατευτούν οι καταναλωτές απέναντι σε αθέμητες πρακτικές των συμβάσεων και να προσφέρεται προστασία παρόμοια με, αυτού, με αυτήν στους, ε, που προσφέρεται στους επιβάτες οι οποίοι αγοράζουν πακέτα ε, ταξιδιών και για παράδειγμα σε ορισμένε περιπτώσεις μετά πτωχεύει η εταιρεία. Τώρα, οι διαδικασίες θα πρέπει να είναι αποδοτικές και ευπρόσιτες. Επίσης και απαρβάνομα λέει ότι τα δικαιώματα των επιβατών είναι ουσιώδους σημασίας και είναι εν τέλει δικαιώματα καταναλωτών και γι' αυτό θεωρεί ότι ο ρόλος της παρόντα Επιτροπή σε οποιαδήποτε μελλοντική αναθεώρηση της ε, νομοθεσία θα πρέπει να ληφθεί υπόψη αφού άλλωστε ε, πρόκειται για προστασία καταναλωτών εν τέλει. Ε, αυτά ευχαριστώ πολύ και αποχωρώ για να πάω στην ραδιοφωνική μου συνέντευξη. Τι κρίμα που δεν μπορούμε να ακούσουμε την συνέντευξή σας με τον κύριο Ντιγιόν. Η κυρία Χέντ Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τον εισηγητή για την εξαιρετική του συνεργασία ε, κατά τη σύνταξη αυτού του εγγράφου. Πρόκειται για ένα εξαιρετικό έγγραφο παρότι έχω υποβάλει πολλές τροπολογίες τις οποίες θα λάβετε εν ευθέτω χρόνο. Συμφωνώ απολύτως με τον εισηγητή για το ζήτημα του ότι τα δικαιώματα των επιβατών είναι, με την εισηγήτρια για το ότι τα δικαιώματα επιβατών είναι δικαιώματα καταναλωτών και αυτό πρέπει να το επαναλαμβάνουμε. Θα πρέπει ο Πρόεδρος να το λάβει υπόψη στο αυτό το ζήτημα για να συνεχίσουμε τις εργασίες μας στο μέλλον σε αυτό το τομέα. Θα πρέπει να μοιραστούν να μοιραστούμε ευθύνε. Δηλαδή, η Επιτροπή Εσωτερική Αγορά θα πρέπει να συμμετέχει, διότι πρόκειται για ε, ζήτημα προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Ε, είναι πολύ ενθαρρυντικό που βλέπουμε να προκύπτει αυτό το ζήτημα. Ε, Εμεί τα μέλη του Κοινοβουλίου ταξιδεύουμε πολύ. Τρέχουμε την Ευρώπη δύο-τρει φορέ την εβδομάδα. Εγώ συχνά έχω προβλήματα με πτήσει που ακυρώνονται ή καθυστερούν. Επίση, ταξιδεύω πολύ συχνά με τρένο μεταξύ Δανία και Σουηδία και αυτό πολλέ φορέ παρουσιάζει προβλήματα όταν έχουμε δύο κράτη-μέλη που εμπλέκονται σε μια υπόθεση. Όπως είπα λοιπόν θα υποβαλώ αρκετά ε, προσθήκες και τροπολογίες για την γνωμοδότηση. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να επιλέξουμε τόσο πολύ κανονισμό. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε μάλλον ότι οι καταναλωτές θα έχουν πρόσβαση σε ένα ελάχιστο σύνολο καλά καθορισμένων κανόνων. Χρειαζόμαστε λοιπόν ελάχιστους κανόνες οι οποίοι θα σεβούνται τις αρχές ε, των δικαιωματών των επιβατών. Συγκεκριμένα μέτρα θα πρέπει να προταθούν για κάθε τομέα των μεταφορών. Είναι σημαντικό κάθε κράτος μέλος να έχει καλύτερη ε, προστασία των καταναλωτών εφόσον το επιθυμεί. Αυτό είναι κάτι που έχουμε εμείς εγείρει ε, σοσιαλδημοκράτες τώρα στο δικό μας τομέα αρμοδιοτήτων για τα δικαιώματα και την προστασία των καταναλωτών είναι σημαντικό να έχουμε κατάλληλα συστήματα για την ε, ε, αποζημίωση σε περίπτωση καθυστερημένων πτήσεων ή ακύρωσης πτήσεων. Θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι παρέχονται επαρκείς πληροφορίες ώστε οι υπηρεσίε παροχή υπηρεσιών, οι ιστοσελίδες ε, να είναι προσβάσιμες και σαφείς όσον αφορά αυτά τα δικαιώματα. Τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος με τα μέσα κοινωνική δικτύωσης, τα smartphone και όλα αυτά. Συνεπώς πιστεύω ότι δεν είναι δύσκολο να υπάρχει εύκολη πρόσβαση στα δικαιώματα των επιβατών όταν αυτό είναι απαραίτητο. Επίσης ε, χρειάζεται να δούμε τι θα κάνουμε με τους ε, επιβάτες μειωμένης κινητικότητα. Χρειάζεται να διασφαλίσουμε ότι θα είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες σε αυτά τα άτομα υπό τη σωστή μορφή. Αυτή η γνωμοδότηση βασίζεται σε μια εκθέση πρωτοβουλίας που μπορεί να οδηγήσει στο μέλλον σε νομοθεσία. Θα πρέπει λοιπόν να μελετήσουμε πιο πολύ πώς μπορούμε να απλοποιήσουμε την εμπειρία των καταναλωτών όταν κάνουν κρατήσεις πτήσεων μέσα στην Ευρώπη. Όταν θέλει τώρα να κάνει μια κράτηση σε τρένο από το Καλμάρ στη Σουηδία όπου μένω εγώ μέχρι το Στρασβούργο πρέπει να περάσει κανεί από πολλέ συνδρομικέ επιχειρήσει, εταιρείε, να επικοινωνήσει με όλε αυτέ, Αυτό είναι κρίμα. Πρέπει να μπορούμε να ταξιδεύουμε όσο μπορούμε περισσότερο στην Ευρώπη και με τρένα και με λεωφορεία όπω κάνουμε και με τι πτήσει. Πρέπει να εξετάσουμε λοιπόν όλα αυτά τα ζητήματα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Τούν. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ την εισηγήτρια. Πιστεύω ότι τα σημεία που αναφέρετε είναι πολύ ακριβή και πολύ σημαντική και όσον αφορά τις προτεραιότητες ένας απλός κανονισμός που να αναφέρει σαφή δικαιώματα για τους καταναλωτές, ισχυρή επιβολή και ούτω καθεξής. Έχω δύο-τρία σημεία τα οποία θα σας αναφέρω και τα οποία θα θέλαμε να προσθεθούν και θα τα αναφέρουμε στις τροπολογίες μας. Το ένα αφορά τη διαλειτουργικότητα. Έχετε κάτι εσείς για αυτό το θέμα και αναφέρθηκε από την Head. Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι θα υπάρχει συνοχή όσον αφορά τα δικαιώματα και ότι αυτό είναι ευθυγραμμισμένο σε υψηλό επίπεδο όταν ας πούμε αλλάζουν τρένο ή πτήσεις ή καταναλωτές είναι το υψηλότερο επίπεδο προστασίας που μπορούμε να παρέχουμε δεύτερον συμφωνώ πάρα πολύ με όσα είπε η πτησεις η καταναλωτες ειναι το υψηλοτερο επιπεδο προστασία που μπορουμε να Χέντ για τους ανθρώπους μειωμένης κινητικότητας τους ανθρώπους με αναπηρία θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι έχουν πρόσβαση όχι μόνο στις υπηρεσίες αλλά και στις πληροφορίες έγκαιρα το τελευταίο που θα ήθελα να αναφέρω είναι κάτι το οποίο δεν είμαι ακόμα βέβαιη ότι θα υποβάλουμε ω τροπολογία αλλά θα ήθελα να το επισημάνω. Αφετηρία μου θα αποτελέσει μια πολύ συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ ευρύτερο. Ακούσαμε από την Κομισιόν ότι περισσότερα, τα περισσότερα παράπονα αφορούν τον τομέα των μεταφορών. Υπήρξε μια περίπτωση στα δανέζικα μέσα ενημέρωση, τα οποία και μου ζητήθηκε να αντιδράσω. Και εγώ δυσκολεύτηκα να απαντήσω. Δανό πολίτη που ταξίδευε με Ισπανό φίλο από τη Δανία προ την Ισπανία και μετά έπρεπε να φύγει προ την Λατινική Αμερική. Με, συγγνώμη, Ισπανική εταιρεία. Καθυστέρησε λοιπόν, έχασε το αεροπλάνο προ την Νότια Αμερική. Δανό πολίτη ταξίδι από Δανία προ Ισπανία και μετά προ Λατινική Αμερική. Και έτσι όπω έχουν τα πράγματα και η νομοθεσία σήμερα, έχει δικαιώματα για αποζημίωση. Υπέβαλε παράπονο, του αναγνώρισε η Ισπανική Αρχή ότι έχει δικαίωμα να λάβει κάποια χρηματική αποζημίωση και κάτι άλλο. Ωστόσο, η Ισπανική εταιρεία δεν τον αποζημίωσε ποτέ. Παρότι η Ισπανική αρχή το ζήτησε, δεν έλαβε ποτέ χρήματα. Όταν επέστρεψε λοιπόν, είπε: Ακόμα δεν έχω λάβει τίποτα. Το ερώτημα λοιπόν είναι τι εργαλεία έχουμε στη διάθεσή μας. Έχουμε καθόλου εργαλεία για τις εταιρείε που δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες. Ακόμη και αφού έχει γίνει μια διαμαρτυρία και αυτή έχει εγκριθεί, σκεφτόμουν λοιπόν ότι Φυσικά έχουμε ε, την ε, δυνατότητες διασυνοριακής επιλύσης διαφορών, τη διασυνοριακή επιβολή, αλλά αυτός μου είπε είναι εξαιρετικά περίπλοκο να, να, καταφύγω στα δικαστήρια στην Ισπανία. Δεν έχω τους απαραίτητους πόρους. Κόστιζε περίπου 2.000 ευρώ και στο τέλος το παράτησε. Και δεν έλαβε ποτέ καμία αποζημίωση. Αυτό ουσιαστικά ζημιώνει την επιβολή μεταξύ των, μεταξύ των συνόρων. Θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε παραπάνω, γιατί φυσικά δεν πρόκειται για τη μόνη περίπτωση. Ένα άλλο σημαντικό σημείο. Αν δείτε το βαθμολόγιο των καταναλωτών, 45% από αυτούς που έχουν προβλήματα δεν καταθέσανε παράπονο γιατί ήταν πάρα πολύ πολύπλοκο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο κύριος Μπιέλ δεν έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχουμε αναφέρει πολλές φορές τα θέματα των δικαιωμάτων των επιβατών και στην προηγούμενη μας γνωμοδότηση σε σχέση με το βαθμολόγιο. Δεν είναι η η Επιτροπή η οποία ασχολείται με τα θέματα αυτά και Επιτροπή Μεταφορών και χαίρομαι για το γεγονός αυτό. Είναι γεγονός όμως ότι πολλές φορές στην Ευρώπη έχουμε καταστάσεις όπου ενώπιον ενός προβλήματος δεν ξέρει ο καταναλωτής πού να πάει και πώς να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Πολλές φορές λοιπόν δεν ξέρουν τα δικαιώματά τους και δεν ξέρουν πώς να βρουν θεραπεία στα προβλήματά τους. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν την κυρία Πιετικάινεν και χαίρομαι που υπογραμμίζει το γεγονός ότι τα δικαιώματα των επιβατών είναι δικαιώματα καταναλωτών και πρέπει να εφαρμόζεται πλήρως η προστασία αυτή. Είναι απαραίτητο να υπάρξει μια αποτελεσματική εφαρμογή αυτών των δικαιωμάτων και συμφωνώ με το σύνολο των προτάσεων που βρίσκονται σε αυτήν την πρόταση. Κάπου που δεν συμφωνώ απόλυτα είναι το σημείο 3 που λέει ότι πρέπει να έχουν ίση προστασία οι καταναλωτές ανεξάρτητα από τον τρόπο μεταφοράς. Ναι, να είναι αποτελεσματική, αλλά αν μπορεί να είναι ίση, αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να εξαρτάται από το είδος μεταφοράς. Δεν μπορούν οι ίδιοι, η ίδια προστασία να την χάνει εγγύησης από όλους τους τρόπους μεταφοράς, γιατί αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πολλά περισσότερα προβλήματα παρά πλέον εκτήματα. Νομίζω λοιπόν ότι κάθε ειδική μορφή μεταφοράς πρέπει να αντιμετωπίζεται διαφορετικά. Δεν μπορούμε παραγωγός χάρη <clears throat> μια μεταφορά με λεωφορείο μικρής απόστασης να έχει την ίδια προστασία με μία μεταφορά από αεροπλάνο σε μεγάλες αποστάσεις. Επομένως, θα πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχουν και ειδικέ αυτές πτυχές και χαίρομαι παρόλα αυτά για την ύπαρξη αυτής της, ε, αυτής της ε, γνωμοδότησης. Και ο κύριος Σφάμπ νομίζω είναι ο άλλος μονάχα ο οποίος έχει να κάνει κάποιο σχόλιο και ο κύριος Κόλσον νομίζω είναι εδώ από την ε, Γενική Διεύθυνση MOVE. Θα του δώσω το λόγο αμέσως. ΣΦΑΠ πρώτα. Σας ευχαριστώ. Πρώτα να ευχαριστήσω για την εισηγήτρια για αυτήν την ολοκληρωμένη ολοκληρωμένο σχέδιο όπως συζητήσαμε και με το βαρόμετρο των καταναλωτών, σημαντικό είναι να ενισχυθεί το ενιαίο των δικαιωμάτων. Ωστόσο, συμφωνώ και με τα κριτικά σχόλια του κ. Μπίλαν, διότι για μένα δεν είναι πολύ σαφές ποια υποτίθεται θα είναι τα 10 δικαιώματα των επιβατών που θα πρέπει να ισχύουν και να εφαρμόζονται ε, ταυτόχρονα ή με τον ίδιο τρόπο σε διαφορετικούς τρόπους μεταφορών, όπου ο κ. Μπίλαν, εγώ βλέπω οι διαφορετικοί τρόποι μεταφορών να αντιμετωπίζουν ή να προκύπτουν σε αυτούς διαφορετικά προβλήματα. Το ίδιο όπως είπε και η κυρία Τούρουνεν προηγουμένως, ότι δηλαδή η εφαρμογή των όσων ήδη διαθέτουμε είναι μεγάλο πρόβλημα. Και εγώ είχα μια παρόμοια περίπτωση στην Ισπανία. Υπάρχουν μεν ξεκάθαροι κανόνες, υπήρξε καθυστέρηση άνω των τριών ώρων, και έτσι προκύπτουν συγκεκριμένα δικαιώματα, ωστόσο δεν υπάρχει μια απλή διαδικασία που να οδηγεί σε αποτελέσματα. Εδώ λοιπόν με ενδιαφέρει ιδίω η εφαρμογή, η εφαρμογή των δικαιωμάτων αυτών, η υλοποίηση των δικαιωμάτων αυτών. Αυτό θα πρέπει να είναι το κυριότερο, το κυρίαρχο στοιχείο που θα πρέπει να ενισχύσουμε. Ευχαριστώ όλες και όλους για τα χρήσιμα σχόλιά σας και θα δώσω το λόγο σύντομα, αν συμφωνείτε, στον κύριο Κόλσον, διότι πολύ χρόνο δεν έχουμε. Αν θέλετε θα σχολιάσετε για ορισμένα από τα όσα ακούσαμε και να μας ενημερώσετε για το πού βρισκόμαστε για ορισμένες από τις ε, πρωτοβουλίες της Επιτροπής Μεταφορών. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την κυρία Πετικάινεν ε, για το σχέδιο έκθεσής της που για εμάς ε, αντιστοιχεί στα σημαντικότερα σημεία που θα πρέπει να επισημανθούν για αυτές τις περιπτώσεις. Συμφωνούμε απόλυτα με τις περισσότερες παρατηρήσεις που έχει διατυπώσει όσον αφορά τη σπουδαιότητα αυτών των δικαιωμάτων και τη σχεδόν συνταγματικής αξίας τους τις διαφορές μεταξύ των μεθόδων στα κράτη-μέλη, τη σημασία της διαλειτουργικότητας, της σπουδαιότητα των παραπώνων και της σπουδαιότητα των επιβατών Μειωμένη Κινητικότητα. Επιτρέψτε μου ωστόσο να κάνω δύο παρατηρήσεις ε, σε σχέση με ομιλίες που ακούστηκαν και που αντιστοιχούν σε ένα από τα σημεία που περιλαμβάνονται στην έκθεση της κυρίας Πετικάινη. Το πρώτο σημείο όταν μια εθνική αρχή ε, δίνει δίκιο σε έναν επιβάτη και ο αερομετοφορέας στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν εφαρμόζει τη σύσταση της εθνικής αρχής, τι μπορεί να κάνει ο εν λόγω επιβάτης. Όπως έχει σήμερα η νομοθεσία, η δυνατότητα που έχει είναι να προσφύγει ενδεχομένως ε, με μια, μέσω μιας απλοποιημένης διαδικασίας που ήδη υπάρχει. Ωστόσο δεν μπορεί να επιτύχει πραγματικά το αποτέλεσμα που θα έπρεπε να προκύψει από την απόφαση της Εθνικής Αρχής. Αντιθέτως, η Εθνική Αρχή εξακολουθεί να έχει τη δυνατότητα να επιβαλεί πρόστιμο. Είναι σαφές λοιπόν ότι ενώπιον του ενδεχόμενου προστίμου είναι πιθανό ή τουλάχιστον δυνατό ή ο αερομοτοφορέας να προσπαθήσει να βρει μια λύση μαζί με τον επιβάτη ή και να εφαρμόσει πλήρως τη σύσταση της Εθνικής Αρχής. Το σύστημα λοιπόν όπως είναι σήμερα δεν επιτρέπει στην Εθνική Αρχή να επιλύσει συγκεκριμένα το πρόβλημα ενός επιβάτη. Αντιθέτως επιτρέπει την έμεση επιλύσή του μέσω του προστίμου που μπορεί να επιβάλλει. Το δεύτερο σημείο στο οποίο θα ήθελα να επανέλθω και το, στο οποίο αναφέρεται η κυρία Πιέτη Κέιναν και για το οποίο μίλησαν πολλά μέλη όπως ο κύριος Μπιλάν και ο κύριος Σουάμπ είναι το ζήτημα των υπαρχουσών διαφορών μεταξύ τρόπων μεταφοράς εδώ ευνοείται σαφώς ε, και αυτός είναι ο στόχος η σύγκληση μεταξύ των διαφόρων τρόπων μεταφοράς. Συμφωνούμε ότι πράγματι στους τρέχοντες κανονισμούς υπάρχουν διαφορές μεταξύ των διαφορετικών τρόπων μεταφοράς που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν αντιθέτως. Εκτιμάμε ότι η απαραίτητα αναγκαία θα συνεχίσουν να υπάρχουν διαφορές διότι έχουμε διαφορετικούς τρόπους μεταφορών. Συνεπώς πρέπει να καταλήξουμε σε μια σταδιακή σύγκληση η οποία ίσως ε, αυτή τη στιγμή είναι πολύ νωρίς για να έχουμε έναν ενίο κανονισμό. Αυτό ενισχύεται από το γεγονός ότι ορισμένοι κανονισμοί όπως ο κανονισμός ε, στον θαλάσσιο τομέα ή ο κανονισμός ε, για τα πούλμαν και τα λεωφορεία δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ. Δεν έχουμε λοιπόν κανένα σχόλιο, κανένα ιστορικό, κανένα από το αποτέλεσμα για να μπορέσουμε να τα κρίνουμε με ακρίβεια. Για αυτούς τους δύο λόγους λοιπόν, ε, οι διαφορές που ε, υπάρχουν, που πρέπει να υπάρχουν μεταξύ των διαφόρων τρόπων και του εξαιρετικά πρόσφατου χαρακτήρα του δικαίου που δεν έχει τεθεί ακόμα σε ισχύ για άλλους τρόπους μεταφοράς, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να περιμένουμε πριν καταλήξουμε σε ενιαία νομοθεσία. Ωστόσο, θεωρούμε ότι προοδευτικά σταδιακά θα καταλήξουμε σε σύγκληση και συμφωνούμε απόλυτα με αυτό. Το μόνο σημείο που θέλω να αναφέρω όσον αφορά την ερώτηση του κυρίου Προέδρου είναι το γεγονός ότι η Κομισιόν πιθανώς θα προτείνει στο τέλος του φετινού έτους μια αναθεώρηση του κανονισμού για τα δικαιώματα των επιβατών στις αναέριες μεταφορές. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία, ωραία. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Πιετικά είναι, θέλει να συνοψίσει. Να μας πείτε και το χρονοδιάγραμμα. Σας ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους αλλά και την Κομισιόν για τα σχόλιά τους. Ήταν πολύ καλά σχόλια και όταν πρόκειται για το θέμα της ίσης προστασίας αυτό που αναφέρατε ήταν πολύ σωστό. πρέπει να καταλάβουμε και το, το θέμα της αναλογικότητος όταν μιλάμε για μικρές ή μεγάλες αποστάσεις. Όταν πρόκειται για την εναρμόνιση. Να σας πω τώρα ποια είναι τα χρονοδιαγράμματα. Η προθεσμία τροπολογιών είναι η 19η Ιουνίου. Η εξέταση θα γίνει στις 9 Ιουλίου, 10 Ιουλίου θα ψηφίσουμε. Ευχαριστώ. Ωραία, ωραία. Προχωράμε τώρα στο τελευταίο σημείο της ημέρας διάταξης, η έκθεση της κυρίας Κόλεν Λάγκεν για την οδηγία καταναλωτικής πίστης δεν είναι παρούσα σήμερα δυστυχώς, αλλά η κυρία Φερχάιεν θα παρουσιάσει την έκθεση εξ ονόματός της. Έχουμε την κυρία Χριστίνα Ρούσο από την Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς και Καταναλωτών. Να δούμε ποιο άλλο είναι παρόν από τις άλλες πολιτικές ομάδες. κυρία Πέντεργάς δεν είναι εδώ, ο κύριος Μπιζό δεν είναι εδώ, η κυρία Ρούλα δεν είναι εδώ. Εγώ είμαι εδώ όμως ο σκιώδης εισηγητής, είμαι ο μόνος επίσημος σκιώδη εδώ. Ίσως να έρθουν και άλλοι, αλλά ούτως ή άλλως πρέπει να ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση και με μεγάλη χαρά δίνω το λόγο στην κυρία Φερ Χάιεν. Σας μεσώ κύριε Πρόεδρε. Η συγγήτρια δυστυχώ δεν μπορεί να παρουσιάσει την έκθεσή της προσωπικά και γι' αυτό με παρακάλεσε να δώσω τα κύρια στοιχεία της έκθεσής της σήμερα. Πρόκειται για την εφαρμογή της οδηγίας για την καταναλωτική πίστη και η πρόταση αυτή που διατυπώθηκε το 2008 είχε δύο στόχους. Να, να προστατεύσει τους ε, καταναλωτές και να ενισχύσει τη διαμεθοριακή εσωτερική αγορά. Η προστασία γίνεται με την ε, εν μέρη εναρμόνιση του καταναλωτικού δικαίου στην Ευρώπη και επίσης πρέπει να τονίσουμε ότι με τον τρόπο αυτό αυξήθηκε η διαμεθοριακή καταναλωτική πίστη από 2% σε 20% που δείχνει τη σημασία αυτού του νομοθετήματος. Αλλά βέβαια είναι λίγες οι, πιστωτικές, τα, οι τράπεζες και πιστωτικά εργαλεία που εφαρμόζουν τη διαμεθοριακή καταναλωτική πίστη και ούτως ή άλλως δεν ήταν αναδρομική ισχύ αυτού του νομοθετήματος. Ένα επιπλέον πρόβλημα ήταν ο χρόνος εφαρμογής δύο χρόνων, όχι μόνο για τα κράτη-μέλη, αλλά και για τα πιστοτικά ιδρύματα. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ πολύπλοκη και έπρεπε επομένω να εφαρμοστεί σωστά και από τον Εθνικό Νομοθέτη και από τα πιστοτικά ιδρύματα και επομένω τα δύο χρόνια δεν έφτασαν. Μας ζητά λοιπόν η συγγήτρια να σκεφτούμε καλύτερα για το μέλλον ώστε να έχουμε ένα χρονικό διάστημα εφαρμογής τριών ετών για ένα τόσο πολύπλοκο νομοθέτημα, για να έχουμε ικανοποιητική εφαρμογή. Υπάρχουν ορισμένα στοιχεία τώρα που θέτουν ένα αμφιβόλο την οδηγία. Παραδείγματο χάρη, το πρότυπο έγγραφο πληροφορίας για την καταναλωτική πίστη, το οποίο έχει επικριθεί ως ιδιαίτερα εκτενές και δυσνόητο. Επίσης, ο υπολογισμός του ε, ετησίου ε, επιτοκίου. Δεν υπάρχει ένας υπολογισμός ο οποίος να, δεν υπάρχουν οι κανόνες υπολογισμού οι οποίοι είναι ταυτόσιμοι. Και τρίτον, ο, η προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων από τον καταναλωτή. Και εδώ υπήρξαν πολλά προβλήματα για να κατανοήσουμε πότε ακριβώς αρχίζει να τρέχει αυτή η προθεσμία. Υπάρχει αβεβαιότητα. Αν ξεκινά από την πρώτη επαφή ή μόνο από την υπογραφή της ε, σύμβασης. Επίσης, επειδή υπάρχουν προβλήματα με την εφαρμογή, η Κομισιόν έχει κάνει μια έρευνα με τη βοήθεια ιστοσελίδων οργανώσεων καταναλωτών. Από όλα αυτά λοιπόν μπορεί κανείς να καταλήξει ότι η οδηγία είναι ένα σημαντικό εγχείρημα για την προστασία των καταναλωτών, αλλά η Κομισιόν θα πρέπει να ελέγξει καλύτερα τα στοιχεία αυτά και ιδίως τα στοιχεία της εφαρμογής στα κράτη-μέλη και να δοθεί επαρκής χρόνος να υπάρξει συλλογή εμπειριών, να υπάρξει πλήρης εφαρμογή και ιδιαίτερα να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα αυτού του μέτρου σε διαμεθαμεριακό επίπεδο και έτσι θα μπορούσε να υπάρξει μια σειρά από που θα αυξήσουν την αποτελεσματικότητα αυτού του εργαλείου για το μέλλον, για ουσιαστικές αλλαγές είναι πάρα πολύ νωρί βέβαια όταν πρόκειται για ένα τόσο μεγάλο, τόσο πολύπλοκο ε, νομοθέτημα. Ευχαριστώ. Ε, thank Σας ευχαριστώ λέει και ο Πρόεδρος. Ως μόνος σκιώδης θα κάνω μερικά σχόλια και να δούμε αν κάποιος άλλος συνάδελφος θέλει να λάβει το λόγο. Πιστεύω καταρχήν ότι οι παρατηρήσεις της κυρίας Κόλεν Λάγκεν είναι ιδιαίτερα χρήσιμες και εστιάζονται πραγματικά στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Είναι εκδηλώ ότι αυτή η οδηγία ήταν κάπως βραδιφλεγής. Πολλοί από εμά που την έχουμε παρακολουθήσει από την αρχή, όπως και εγώ ο ίδιος, ξέρουμε ότι ξεκίνησε αυτή η διαδικασία πριν από περίπου 13 χρόνια και είχαμε μακρές συζητήσεις για τα θέματα εναρμόνισης και της σκοπιμότητας της ε, εναρμόνισης. Και υπήρχε τότε μια ισχυρή άποψη στο Συμβούλιο αλλά και στο Κοινοβούλιο ότι είναι τόσο διαφορετικές οι αγορές καταναλωτικές πίστης στα κράτη-μέλη, που η αξία μιας πλήρως εναρμονισμένης οδηγίας θα ήταν, για οδηγίες για πλήρη εναρμόνιση καλύτερα, θα ήταν πολύ περιορισμένη. Η κυρία Κόλεν Λάγκεν έχει αναφερθεί στο επίπεδο των διαμεθοριακών συναλλαγών καταναλωτικής πίστης που παραμένει ακόμα σε χαμηλό επίπεδο. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν σημαντικές πτυχές προστασίας των καταναλωτών, οι οποίες έχουν τύχη εναρμόνισης. Και τώρα η έρευνα SWEEP που ανέφερε η κυρία Κόλεν Λάγκε δείχνει ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά σε σχέση με τις παρεχόμενες πληροφορίες που είναι ένα από τα κύρια πράγματα που μας ενδιαφέρουν και ιδίως η μορφή με την οποία παρουσιάζονται όλα αυτά τα στοιχεία μέσα σε κοιτία και ε, όπως είδαμε και προηγουμένως με την παρουσίαση του βαθμολογίου θα είναι χρήσιμο να δούμε αυτά τα συγκεκριμένα στοιχεία και το πώς συνδέονται με τα παράπονα των καταναλωτών. Κάτι άλλο το οποίο καλύπτει η κυρία Κόλεν Λάγκεν και το οποίο θα ήταν ενδιαφέρον να το ε, αντιμετωπίσουμε με τροπολογίες είναι η διαθεσιμότητα στοιχείων σε διαμεθοριακό επίπεδο για το, τη βαθμολογία που δίδουν οι καταναλωτές. Γιατί αυτός είναι και ο τρόπος που χρησιμοποιούν οι καταναλωτές για να, δουν τι δυνατότητες τους δίνουν μεγαλύτερη φερεγγιότητα. Και υπάρχουν αντιμαχόμενες απόψεις σε σχέση με αυτή τη βαθμολογία. Κάτι το οποίο ήθελε να επιτύχει η οδηγία αυτή είναι να ανοίξουν αυτές οι βάσεις δεδομένων σε διαμεθοριακό επίπεδο για όλους τους διακινούμενους και μη πολίτες, αλλά φυσικά και αυτό συνάπτεται με πάρα πολλά θέματα. Νομίζω ότι σωστά η κυρία Κόλεν Λάγκεν αναφέρεται στο θέμα των συστημάτων πληρωμής, όπου υπήρχαν διαφορετικές προτάσεις, παραμένει ένας πολύπλοκος χώρος. Έχουμε συμφωνήσει ήδη με την Κομισιόν σε επίπεδο επιτροπολογίας να αλλάξουμε το τον τρόπο υπολογισμού του επιτοκίου σε ετήσια βάση, αλλά αυτό είναι κάπως δύσκολο για τους καταναλωτές να γίνει κατανοητό και το τελευταίο σημείο που θέλω να θίξω σήμερα, γιατί θα επανέλθουμε, είναι το θέμα του πεδίου εφαρμογής. Πήγαμε πριν από δύο χρόνια στην ε, Σουηδία, κατά τη διάρκεια της Προεδρίας Σουηδίας, και το Κοινοβούλιο της Σουηδίας αναφέρθηκε στα λεγόμενα δάνεια με SMS. Εμείς από ό,τι τους είπαμε, θεωρήσαμε ότι θα μπορούσε η κυβέρνηση Σουηδίας να εφαρμόσει αυτό το νομοθέτημα και σε τέτοιου είδους συναλλαγές. Και η κυρία Κόλε Λάγκεν αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο ορισμένα κράτη-μέλη έχουν συμπεριλάβει και υποθήκες, στεγαστικές υποθήκες. Και θα έπρεπε να δούμε και πάλι τι θα γίνει με την πρόταση για τα στεγαστικά δάνεια της Κομισιόν, όπου πολλοί ήταν σκεπτικιστές, αλλά όπου και η δική μας θέση ήταν να μεταφέρουμε πολλές ε, διατάξεις και πρόνοιες της ε, οδηγίας για την καταναλωτική πίστη σε σχέση με την παροχή πληροφοριών πριν από τη σύναψη της σύμβασης για να έχουμε μία κάποια συνεκτικότητα. Γνωρίζω ότι ο εισηγητή τη Επιτροπή ΕΚΟΝ ήταν λίγο πιο φιλόδοξο όσον αφορά την ε, ε, προστασία των καταναλωτών. Θα δούμε ποια θα είναι τα δικά του σχόλια. Θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε κατά πόσο η κυρία Ρίτερ εκ μέρου τη Επιτροπή ε, συμφωνεί με την κατεύθυνση που επιλέγει η κυρία Δηλαδή θεωρεί ότι δεν υπάρχει μεγάλη ανάγκη αυτή τη στιγμή για σημαντική τροπολογία των διατάξεων της υπάρξης οδηγίας. Θα πρέπει μάλλον να επικεντρωθούμε στο να διασφαλίσουμε τη σωστή της υλοποίηση και να αντιμετωπίσουμε τα όποια ζητήματα υλοποίηση που προκύπτουν από την υπάρχουσα οδηγία αντί να προτείνουμε ε, ριζική μεταρρύθμιση. Επίση, το να συμβουλέψουμε ειδικότερα τα κράτη-μέλη ενδεχομένω το πώ μπορούν να χρησιμοποιήσουν πιο αποτελεσματικά την οδηγία από όσο πράττουν σήμερα. Εφόσον συμφωνούμε με την Κομισιόν, αυτή είναι, αυτό είναι το σκεπτικό για μια έκθεση πρωτοβουλίας ε, πριν λάβουμε την πρότασή σας. Γνωρίζω ότι έχετε προβεί και σε πιο εκτενείς διαβουλεύσεις και θα ήθελα να μάθω το χρονοδιάγραμμά σας ώστε να μπορούμε να προγραμματίσουμε κι εμείς ε, πώς θα προχωρήσουμε στο μέλλον. Κάποιος άλλος. Η Χριστίνα, παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε την κυρία Φερχάιεν για την παρέμβασή της για την έκθεση Colin Langen. Με την ερώτησή σας ε, με διευκολύνεται. Μπορώ να σας πω απλά ότι συμφωνούμε με την κατεύθυνση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτή την έκθεση. Πιστεύουμε ότι πρόκειται για μια σημαντική οδηγία και θεωρούμε ότι το ζήτημα εδώ είναι να διασφαλιστεί, το πρωταρχικό ζήτημα είναι να διασφαλιστεί η σωστή της υλοποίηση όπως αναφέρεται στην έκθεση και όπως αναφέρθηκε και από εσάς ε, κατά τις διάφορες παρεμβάσεις ε, παρατηρήθηκαν κάποιες δυσκολίες στα κράτη-μέλη όσον αφορά την υλοποίηση αυτής της οδηγίας. Ορισμένες από αυτές τις δυσκολίες προσπαθήσαμε να τις αντιμετωπίσουμε με τροποποιήσεις ε, των παραρτημάτων αυτής της οδηγίας τροποποιώντας ε, κάποια ε, υπολογισμούς ε, του APR όπως αναφέρατε πολύ σωστά και επίσης παρήχαμε κάποιες κατευθυντήριες γραμμές στα κράτη-μέλη για την υλοποίηση της οδηγίας κατευθυντήριες γραμμές που Επίσης εστάλησαν και στη γραμματεία της παρούσας επιτροπής αν δεν κάνω λάθος εάν αυτό δεν έχει γίνει φυσικά και θα τη στείλουμε για εμάς είναι πολύ σημαντικό πολύ σημαντική η κατεύθυνση που επιλέγετε. Συμφωνούμε απόλυτα μαζί σα, Πρέπει να υποστηρίξουμε τα κράτη-μέλη όσον αφορά τον τρόπο υλοποίηση αυτής της οδηγίας. Αλλά υπάρχει και άλλο ένα σημείο από αυτά που είπατε, για το, στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ. Είναι πολύ σημαντικό οι διατάξεις της οδηγίας να γίνουν γνωστές στους καταναλωτές, να υπάρξει ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των καταναλωτών όσον αφορά τα δικαιώματα που αποκτούν με αυτή την οδηγία. Γι' αυτό το λόγο Προσπαθούμε να δούμε κατά πόσο θα ήταν δυνατό να οργανώσουμε μια ενημερωτική εκστρατεία για την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών όσον αφορά τα δικαιώματά τους ε, υπό την οδηγία καταναλωτικής πίστης. Τώρα η ερώτηση κατά πόσο μπορούμε να επεκτείνουμε τις διατάξεις και στα δάνεια προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στα στεγαστικά δάνεια, ναι θα είναι δυνατόν. Ε, τώρα όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, δεν το είπατε, αλλά υπάρχει μέσα στην έκθεση. Αυτή τη στιγμή γίνεται μια μελέτη αγοράς για τις επιπτώσεις αυτής της οδηγίας. Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης αναμένονται για τα τέλη του έτους. Ταυτόχρονα ολοκληρώνουμε τους ελέγχους μεταφοράς, δηλαδή πώς τα κράτη-μέλη υλοποίησαν αυτές τις διατάξεις. Έχουμε καθυστερήσει σε αυτούς τους ελέγχους μεταφοράς, όχι επειδή εμείς καθυστερήσαμε, αλλά επειδή οι μεταφορές στο εθνικά δίκαια έγιναν καθυστερημένα. Ε, οκτώ μονοκράτη μέλη έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία. Πιστεύουμε ότι θα έχουμε μια πλήρη εικόνα μέχρι τα τέλη του έτους. Στη συνέχεια θα συντάξουμε, όπως προβλέπετε, μια έκθεση το 2013. Έκθεση σε σχέση με τον τρόπο υλοποίησης της οδηγίας για την καταναλωτική πίστη. Και τότε θα δούμε κατά πόσο υπάρχει ανάγκη αναθεώρησης ορισμένων διατάξεων ξεκινάμε ε, θεωρώντας δεδομένο ότι αυτό που θέλουμε είναι να διασφαλίσουμε τη σωστή υλοποίηση παρά την αναθεώρηση της οδηγίας. Ε, ελπίζω να ήμουν σαφής. Ευχαριστούμε πολύ για το ενδιαφέρον σας και θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μας σε αυτό το φάκελο. Ευχαριστώ. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, χαίρομαι ιδιαίτερα που ε, ακολουθούμε την ίδια κατεύθυνση. Φυσικά θα πρέπει να ακούσουμε και τις απόψεις των υπολείπων πολιτικών ομάδων πριν οριστικοποιήσουμε τη θέση μας. Έχετε άλλα μηνύματα κύριε Βερχέβιν ή απλά να συνοψίσω. Συνοψίζω λοιπόν. Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, 30 Ιουνίου για τροπολογίες θα τις μελετήσουμε 17 και 18 Σεπτεμβρίου, συμβιβασμοί 10 Οκτωβρίου και ψηφοφορία στην 11η Οκτωβρίου. Αυτό μας δίνει αρκετό χρόνο για να συντονιστούμε με τις διαδικασίες της Κομισιόν και έτσι θα μπορέσουμε να λάβουμε και αρκετά σχόλια από τις πολιτικές ομάδες. Ε, ευχαριστούμε πολύ την κυρία Κολίν Λάγκεν, εν απουσία της βέβαια. Έτσι κλείνουν οι εργασίες μας για σήμερα. Τελειώνουμε νωρίτερα. Ευχαριστώ συνήθω τους διερμηνεί. Είναι λίγο παράξενη αυτή η αίθουσα για μια συνεδρία επιτροπή, ε, αλλά τουλάχιστον έχει περισσότερο φως, ε, φυσικό. Θα ήθελα να υπενθυμίσω τα μέλη, στα μέλη δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, ότι στην Ολομέλεια της επόμενης εβδομάδας, την Τετάρτη το απόγευμα, θα γίνει μια πολύ σημαντική συζήτηση με τον κύριο Μισελ Μπαρνιέ, τον επίτροπο Μισελ Μπαρνιέ, για τρία σημαντικά ζητήματα. Την νέα του έκθεση για την υλοποίηση της οδηγίας για τις υπηρεσίες, την έκθεσή του για τη διακυβέρνηση στην ενιαία αγορά και επίσης τις προτάσεις για την επόμενη φάση του Single Market Act, Single Market Act 2. Η Επιτροπή μας έχει υποβάλει ένα ψήφισμα που ψηφίστηκε στην Επιτροπή την περασμένη εβδομάδα και που θα συζητηθεί φυσικά από τις πολιτικές ομάδες. Ελπίζω ότι και τα μέλη της Επιτροπής θα συμμετέχουν στη συζήτηση. Η επόμενη συνεδρίασή μας είναι στις 20 και 21 Ιουνίου από 9 το πρωί και τις δύο ημέρες πλήρης ε, συνεδριάσεις όπου θα ψηφίσουμε σε μεγάλο αριθμό, για μεγάλο αριθμό προτάσεων που έχουμε μελετήσει κατά τη διάρκεια του έτους. Ε, προσδοκώ να σας ε, συναντήσω τότε και ευχαριστούμε και το κοινό που μας παρακολουθεί ε, μέσω διαδικτύου πέρα στη συνεδρία. Ευχαριστώ πολύ.